nutzen, was ich jetzt auch benutze, Entschuldigung. Also immer das linke Mikrofon benutzen, falls Sie reden und ansonsten daran denken, dass να χρησιμοποιείτε παρακαλώ το μικρόφωνο όταν ε, έχετε το λόγο και θέλετε να μιλήσετε και να μην ξεχνάτε ότι ε, μπορούν να μας δουν από το διαδίκτυο. Η μερίσια διάταξη. Είναι κανείς κατά? Όχι. Σημείο έγκριση των πρακτικών. Τάχετε τα πρακτικά. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτά ή αν έχετε προβλήματα. Άμα έχετε ήδη από τώρα προβλήματα, πείτε τα από τώρα. Δεν βλέπω όμως κανέναν. Στα βουλγαρικά, τσεχικά, ε, λιθουανικά, εσθονικά μαλτέζικα, ελωτεωνικά, πορτογαλικά, σλοβενικά δεν έχουμε διερμηνία, αλλά οι Ολλανδοί μπορούν να μιλήσουν στα Ολλανδικά. Δεν υπάρχει στα Ολλανδικά διερμηνία. Έχετε και μία έκθεση για το ταξίδι που έκανε μία αντιπροσωπεία μας στο Άρχος. Θα το στείλουμε και στην Προεδρία, στον Πρόεδρο, στο Προεδρείο. Ε, κάποιοι θα πάνε στο Πλόφτιφ αύριο. Δεν είναι και εδώ στη γωνία, πρέπει να φύγουμε νωρίτερα από την αντιπροσωπή, Από τις 10 η ώρα θα με αντικαταστήσει εδώ η κυρία Τρίπελ. Πάμε στο σημείο 4. Το πρώτο επί της ουσίας είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό. Ένα από τα σημαντικά προγράμματα είναι πολιετές και πρέπει να ασχοληθούμε και να το αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Είχαμε μία ακρόαση φέτος, αν θυμάστε, τον Απρίλιο. Είχαμε την ακρόαση και ακούσαμε από όλου που ήταν εκεί ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του τομέα του πολιτιστικού από τη μια και του τομέα των μέσων ενημέρωσης ε, ελήφθησαν υπόψη και πρέπει να συνεχιστούν να λαμβάνονται υπόψη. Ε, έχουμε το, την ονομασία μέσα και όταν ε, αναφέρεται οριζόντια και κάθετα για την Ευρώπη είναι και ο μη κερδοσκοπικός τομέας που προστίθεται εδώ και το εμπορικό, τα εμπορικά προγράμματα. Η Σίλβια Κώστα, η συγγήτριά μας, υπέβαλε ένα έγγραφο εργασίας και θα μας το παρουσιάσει και θα συζητήσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, προσπάθησε να ε, συνεργαστεί καλά και με τους σκιώδεις Βέβαια, αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τότε πρέπει δημοκρατικά να ληφθεί μια απόφαση, δεν γίνεται αλλιώς. Όμως θα δούμε στο τέλος της συζήτησης αν χρειάζεται να δοθεί παράταση ή όχι. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στη Σίλβια, όμως, για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ, Σίλβια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε στην εισαγωγή σας, Προσπάθησα την έκθεση μου να λάβω υπόψη και όσα προέκυψαν από ε, την ακρόαση στην Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά και στις συναντήσεις που είχα με ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και με φορείς, θεσμούς, αλλά και στις ε, συνομιλίες που είχα και με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, συναδέλφους τους Κιώδης, με τους οποίους είχαμε, ελπίζω, μία σημαντική και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και με όσους βεβαίως ε, συνεργάστηκαν μαζί μου και ιδίως ε, τη γραμματεία την οποία ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια. Ξεκινώ με μία σκέψη ουσίας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημιουργική Ευρώπη περιέχει μία σειρά σημείων που πρέπει να δούμε θετικά. Απλά θα σας υπενθυμίσω ε, εντάχει. Όχι μόνο ανάπτυξη αύξηση του προπολογισμού κατά 30% για να φτάσουμε σε 1,8 δισεκατομμύριο τους πόρους για αυτό το τομέα, αλλά και για να ξεκαθαρίσουμε τους τέσσερις προκλήσεις, καθώς ο τομέας ε, που είναι πραγματικά τεράστιος, καθώς περιέχει πάρα πολλά στοιχεία, τομέα του πολιτισμού και περιέχει βεβαίως και τη δημιουργικότητα και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τα μέστα. μέσα. Κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς, παγκοσμιοποίηση και ανταγωνιστικότητα, ψηφιοποίηση και η δύσκολη πρόσβαση ε, στα δάνεια, ιδίω για τι προμεσαίε επιχειρήσει. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που ασπαζόμαστε σε σχέση με όσα προτείνει η Κομισιόν είναι ότι ανοίγει μάλλον το πρόγραμμα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο ε, συμμετεχών στον τομέα του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας καθώς είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την καινοτομία και την ε, βιώσιμη οικονομία και βεβαίως με την πρόσβαση σε δάνεια για την πραγματικότητα. Αυτό είναι βεβαίως κάτι που δέχτηκαν πολύ θετικά και πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι φορείς της μας. Τώρα θέλω να πάω πιο πολύ στις διαφορέ που έχουμε και στις διαφορετικέ επιλογές που προτείνουμε, όπως φαίνεται στην εκθεσή μου, ότι η ενσωμάτωση δεν μπορεί να σημαίνει και μία αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιαίτερων αναγκαίων που έχει ο τομέα τη δημιουργικότητα ε, σε σχέση με το οπτικοστικό τομέα που έχει μια συγκεκριμένη διάρθρωση. Έχει μια βιομηχανία στι πλάτε. και πιο πολύ έχει, αν θέλετε, και την αγορά ως αποδέκτη. Γι' αυτό λέμε το πολύ Δημική Ευρώπη, το πρόγραμμα Δημική Ευρώπη, να αποτελέσει πρόγραμμα πλαίσιο, που θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Πολιτισμός από τη μία, που να περιέχει την πολιτισμό και δημιουργικότητα δηλαδή, και από την άλλη τα μέσα ενημέρωση με προτεραιότητες στόχους. Κριτήρια αξιολόγησης, αποδέκτες, και ε, ειδικά σήματα. Και εδώ ε, η καινοτομία θα είναι και μία ε, διατομιακή διάσταση. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια διαφοροποιημένη κατανομή του κρατικού προπολογισμού. Γι' αυτό αποφάσισα να εντάξω στην εκθεσή μου, όπως βγήκε μάλλον και από τις συζητήσεις που είχαμε, και έναν ορισμό της έννοιας επιμερισμού των πόρων, 55% τουλάχιστον πρώην για το Μέντια, 35% για τον πολιτισμό και 20% ε, το ποσό για ε, τον, ε, τη διατηματική διάσταση. 4% τουλάχιστον για τα διεθνικά μέτρα. Το μέγιστο δυνατό μέσο που θα διατίθεται, όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα, θα παίρνει το 5% του, προπολογισμού. Και σε κάποια περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5% ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν περισσότερα προγράμματα. Προσπάθησα λοιπόν να εξισορροπήσω από τη μία τι αναγκαιότητε, να ορίσουμε τα πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα επαρκέ επίπεδο ευελιξία, ώστε την επόμενη πραγματική περίοδο να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε έναν τομέα που αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές και μεταμορφώνεται ώστε να έχει ένα πιο ισχυρό ρόλο το Κοινοβούλιο στην καθοδήγηση ε, των ετήσιων προγραμμάτων. Επ' αυτή την έννοια, με βάση το άρθρο 290 τη Συνθήκη Λειτουργία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνω το ετήσιο πρόγραμμα να ε, εγκρίνεται με κατευθυντότητες πράξεις που να ορίζουν στόχους αναμενόμενα αποτελέσματα, συνολική χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα. Η πρότασή μου για τους όρους προσχώρησης για προγράμματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για τις υποψήφιες χώρες, χώρες, ε, διαδικασία ένταξη σε χώρες ΕΖΕΣ, Ελβετία και οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια διαβάθμιση της προσβασιμότητας σε αυτά τα κονδύλια. Με βάση την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα καθώς που να λάβουμε υπόψη τους μακρύς χρόνους που χρειάστηκαν για να προσαρμοστούν αυτές οι χώρες, δηλαδή πολλές χώρες χρειάστηκαν ε, μπαίνουν σε διαδικασία πέντε χρόνια για να μπουν σε τη διαδικασία και ο κίνδυνο είναι πολλέ χώρε να μην καταφέρουν καν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματο να έχουν το δικαίωμα να γίνουν δικαιούχοι στο πρόγραμμα Media. Οπότε πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Έπειτα στου ορισμού, να ορίσουμε καλύτερα τους όρους της ψυχαγωγικής πολιτισμού οπιακουστικά μέσα. Έπειτα στον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε τα μουσεία επίσης και ε, επίσης και τη μόδα όπως προβλέπει και η σχετική πράσινη βίβλος. Έπειτα για τους εμπορικούς φορείς. Οι φορείς μάλλον γενικότερα καλύπτουν και τις μη και κερδοσκοπικούς και μη οργανισμούς και ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους μη κερδοσκοπικούς φορείς και να δώσουμε ένα σαφή ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, υπό τους όρους που ε, μας ενδιαφέρουν εδώ για την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Η, κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια ισοποίηση παιδοποιημένη αν θέλετε προσέγγιση καθώς έχει ως γνώμονα μόνο το οικονομικό κέρδος. Με τον κύριο Καβαδά πιστεύω ότι είχαμε και πολλά σημεία ταύτισης εν προκειμένου στην μας και επισημαίνω ε, επίσης ότι ο πολιτισμός σήμερα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και σε εθνικό και περιεθνικό επίπεδο για την τοπική ανάπτυξη, για τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Γι' αυτό μεταξύ λοιπόν των γενικών στόχων του προγράμματος σε περιλαμβάνω την προστασία και την πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ηλική και άλλης, ταυτόχρονα με την προστασία της πολιτισμικής διαφορετικότητας και στήριξη των δημιουργικών επιχειρήσεων. Έπειτα, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο ρόλο στους ίδιους τους φορείς του πολιτισμού, στους ανθρώπους και ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στους νέους, τα παιδιά και τα άτομα ε, σε μειονεκτική θέση και τις ομάδες που επεκρουσαπούνται και τέλος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση και στο εξή. Να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην κυκλοφορία των έργων τέχνη και των γυναικών καλλιτεχνών που πολύ συχνά υποπεκπροσωπούνται ε, ακόμα και στου δημόσιου πολιτιστικού φορεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, μάλλον συγγνώμη την ε, διατομιακή διάσταση του προγράμματο, θα λαμβάνει υπόψη δύο στοιχεία τη νέα, το νέο δημοσιονομικό εργαλείο και τις διαδομικές πολιτικές. Το νέο λοιπόν οικονομικό εργαλείο θα πρέπει, και αυτό το ξεκαθαρίζουμε στην έκθεσή μας, θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, όλους τους ε, πόρους που θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και αυτό θα είναι μια εγγύηση, είναι πολύ αναγκαίο εργαλείο, αλλά δεν ορίζεται σαφώς το πώς θα, γίνει, θα χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός στην πρόταση της Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν διευκρινίζω κάποιες πτυχές που θεωρώ πολύ σημαντικές πράγματα που έφυξαν και εδώ οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Πολιτισμού αλλά και διάφορα διαφοροι διαφορεμένοι φορέ. φορεί. Λοιπόν, δύο-τρία στοιχεία που θέλω να αναφέρω. Λοιπόν, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι φορεί με έδρα στα κράτη-μέλη. Φορέ που έχουν ήδη έχουν μια εμπειρία στο παρελθόν στον τομέα, είναι κάτι που συμμερίζουμε, επί τα μηχανισμοί ελέγχου που θα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθούμε να τη διευκρινίσουμε περαιτέρω και ζήτησα, να δημιουργούνται χαρτοφυλάκια Αυτά τα εργαλεία ευρωπαϊκής εγγύησης θα πρέπει να βοηθούν για την δανειοδότηση των διαφερομένων, ώστε να μπορούν σε εθνικό επίπεδο να δίνονται αυτά τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε επιμέρους οργανώσεις, οργανισμούς, ενώσεις. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χαρτοφυλάκια να είναι ισορροπημένα και να συνοδεύονται και από σχέδια marketing που κάτι που δεν προβλεπόταν στο παρελθόν. Και επίσης διευκρινίσουμε και ποιες θα είναι οι δράσεις που θα πρέπει να έχουν οι διαμεσολαβητές εν προκειμένου που θα αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, έκρινα σκοπό να ξεκαθαρίσουμε τι είδους δάνεια, θα μπορούσαμε να προστάσουμε κι άλλα, αλλά ήθελα να πω εγώ κάποια πράγματα, τι είδους δάνεια εννοούμε. Και καταλήξαμε σε τρία επιλέξιμα δάνεια ε, επενδύσει σε υλικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για άλλα περιουσιακά στοιχεία, εδώ ακριβώς μιλάμε για πνευματική ιδιοκτησία, Και έπειτα, η δεύτερη κατηγορία ε, δανείων είναι η μεταβίβαση επιχειρήσεων, και τα κεφάλαια κίνηση, ε, η προσωρινή χρηματοδότηση, δηλαδή διάφορες μορφές χρηματοδότησης δανείων που θα πρέπει να είναι επιλέξιμες. Καθώς οι γνωστές επιχειρήσει είναι τόσο πολλές και διαφορετικές που απαιτούν ε, μια τέτοια προσέγγιση διαφοροποιημένη. Σε ό,τι αφορά την άλλη διάσταση αυτής ε, της διατομικής συνιστώσας, επειδή ξέρουμε ότι η καρδιά αυτού του προγράμματο είναι να ενθαρρύνει την κυκλοφορία των καλλιτεχνών, των αργοτέχνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ είναι σημαντικό όχι μόνο τα business models, τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα πρέπει να υποστηρίξουμε, αλλά και τα μοντέλα επιχειρηματικότητας, το επιχειρήν που θα έχει σκοπό να δημιουργήσει και νέες συμπράξεις σε δημόσιο-ιδιωτικό τομέα όπως και χρήση όλων των μέσων και ιδιαίτερα τα ψηφιακά μέσα. Ενισχύεται επίσης ε, ο τομέας της παιδείας, η χρήση της ε, ψηφιακή, του ψηφιακού αλφαβητισμού, ο κινηματογράφος, ε, η επαγγελματική κατάρτιση προς αυτή την κατεύθυνση και δίνοντας πρωτεύοντα στην κινητικότητα. Ξέρουμε ότι μεγάλη πρόκληση προκειμένου είναι οι κατάλληλε ε, δεξιότητες, η προσαρμογή των δεξιοτήτων των διαφερομένων. Θέλω να πω ότι συμφωνούμε με αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ο τομέα θα πρέπει να έχει μία σειρά, μάλλον μία δέσμη δεδομένων και δικτών. Αυτό προέκυψε από όλε τι συζητήσει που είχαμε η επιλογή της Επιτροπής, της Κομισιόν, συγγνώμη, αυτό να προβλέπεται σε όλους τους μέρους τομείς και αυτό να γίνεται από, τον, ε, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοστικών Μέσων, θεωρεί ότι είναι μια πρόημη και πρόορη στάση. Τα οπτικοστικά μέσα είναι ένα πολύ σημαντικός επιμέρους τομέας του πολιτισμού, αλλά δεν καλύπτει τα πάντα. και εμείς. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε προσυπογράψει και μία σύμβαση με το Συμβούλιο Σοβαρά σε αυτή την κατεύθυνση που ε, θα πρέπει να ξαναδούμε. Λοιπόν, το παρατηρητήριο θα πρέπει να κρατήσει τι αρμοδιότητε που έχει. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αντιρρήσει. Αλλά αυτό αφορά τα αποκλειστικά μέσα. Από εκεί πέρα η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια μελέτη σκοπιμότητα για το τομέα του πολιτισμού δημιουργικότητα και να μα υποβάλει τα αποτελέσματα τη ε, ε, μελέτη εδώ μέσα σε ένα χρόνο από τη θέση ισχύ του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τα desk Δημιουργική Ευρώπη, να πω ότι προέκυψαν και κάποια ερωτηματικά και από το Συμβούλιο. Δηλαδή, συμμετέχουσε στο πρόγραμμα χώρες να είναι αυτές που θα επιλέξουν το περιεχόμενο. Δηλαδή, α, θα έχουμε ένα desk, ενίοτε για όλη την Ευρώπη ή πολύ περισσότερα. Δεν παίρνω θέση. Έπειτα στο κείμενό μου αναφέρουμε στο ρόλο και τα καθήκοντα του καθενός για την ε, παροχή βοήθειας που θα πρέπει να δίνουν τα desk αυτά, αυτά τα γραφεία αν θέλετε. Αν δημιουργήσουμε ένα δίκτυο τέτοιων γραφείων θα έχουμε και ένα καλύτερο συντονισμό σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πολιτισμού μεταξύ των ε, προτεραιοτήτων δίνουμε έμφαση στα νέα επιχειρησιακά μοντέλα οι δημιουργικέ συμπράξει ω όρο είναι κάτι που όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή γλώσσα, αλλά και την ενεργό συμμετοχή. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή. Σκεφτείτε μόνο τη διάδοση νέων πρακτικών για να συμμετάσχει πιο πολύ το κοινό σε αυτές τις εθνικές συμπράξεις. Σκεφτείτε δηλαδή τι είδου εμπειρίε θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη νύχτα των μουσείων, φεστιβάλ φιλοσοφία και λογοτεχνία, καλλιτεχνικέ διαδρομέ, εφαρμογέ ε, ε, στα θέατρα και στην όπερα. Και βεβαίω το πρόγραμμα πολιτισμός μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τα τοικοστικά μόνο επικουρικά και αν έχει ως σκοπό να υπηρετήσει τους στόχους του προγράμματος πολιτισμός. Έπειτα, για να προωθήσουμε την ε, κυκλοφορία, αν θέλετε, των ε, έργων τέχνης, εδώ θα πρέπει και πάλι να προάγουμε την λογική των φεστιβάλ, αλλά και τις ψηφιακές πλατφόρμες πλατφόρμες με αρχαία ψηφιακά, με ψηφιακές βιβλιοθήκες, ε, πολιτιστικών αγαθών, μετάφρασή τους, επειδή και ο υποτετλισμός, ο μεταγλωτισμός, η μεταγλώτηση συγγνώμη, και η μεταφορά των έργων και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έπειτα συμφωνούμε τη θέση του Συμβουλίου ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ιδιαίτερα τα project των μη κερδοσκοπικών φόρων. Και λίγα λόγια για το πρόγραμμα Media, ότι οι προτεραιότητε και τα μέτρα που ήδη έχουν δει θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Θα πρέπει δηλαδή το πρόγραμμα να παραμείνει αυτόνομο, θα πρέπει να συνεχιστεί να, να προστατεύονται οι καλλιτεχνικοί φορείς και όλοι όσοι ως τώρα συνέβαλαν τα μάλα και κατέστησαν το πρόγραμμα ΜΕΤΙΑ ένα επιτυχές πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να επιτυχθεί μια νέα ισορροπία χρησιμοποιώντας την Αγινέα επιχειρησιακά μοντέλα ώστε να δώσουμε μια νέα αξία στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική ταινία χρησιμοποιώντας βεβαίως και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Μίζωνο σημασία προκειμένου είναι να δώσουμε έμφαση στην παιδεία για τα μέσα, το media literacy και την εκπαίδευση μέσω του κινηματογράφου. Μέσα τώρα που θα βοηθήσουν αυτό είναι η διανομή των κινηματογραφικών έργων στις κινηματογραφικές αίθουσες και ε, η διορυφορική μετάδοση, οι δορυφόροι μπορούν να δώσουν και μία δεύτερη ζωή, αν θέλετε, σε αυτά τα έργα τέχνης, Έπειτα, υποτιτλισμός και μεταγλώτηση. Φυσικά και θα βοηθήσουν την κυκλοφορία των οπιοκουστικών ε, έργων. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στην απόδοση και τη διάδοση όλων αυτών. Πολύ σημαντικό στοιχείο στη συζήτησή μα είναι ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν την συμπληρωματικότητα της Δημιουργικής Ευρώπης με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Συνοχή, ιστορική αγορά, υγεία, νέοι, τα πάντα. Με τα διαφορετικά ταμεία και την έρευνα, όπως επίσης και με την ψηφιακή ατζέντα, γιατί εκεί χρειάζονται καλύτερα συνέργειες. Και τέλος, εύχομαι να υπάρχει συντονισμός με τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση, το πρόγραμμα προβλέπει ότι ένα ανεξάρτητο φορέα θα κάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματο πλαίσιο, αλλά λέω εγώ τώρα, εδώ στην εκθεσή μου, ότι πέρα από του ποσοτικούς δείκτε που εγώ α, ναι, ξέρω ότι αυτό είναι ευαίσθητο ζήτημα, αλλά επειδή μιλάμε για πολιτισμό, να ζητήσουμε την Κομισιόν στις κατά αξιοδότηση, να ορίσει και μία δέσμη ποιοτικών δικτών που θα θέσει υπόψη μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περιπλόκο ε, Αυτέ είναι οι βασικέ επιλογέ. Πρόεδρε, να σταματήσω εδώ. Απλά ήθελα να σας ξεκαθαρίσω το τοπίο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ε, του κοιόδης και με το καλοκαίρι στη μέση δεν ήταν εύκολο να οργανώσουμε τις συναντήσεις μας. Ζητώ συγγνώμη. που δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε και αρκετά συχνά. Πάντω ήταν εξαιρετική συνεργασία με όλου σα και βεβαίω να πω ότι εξ αρχή θα ακούσω με μεγάλη προσοχή ό,τι έχετε να πείτε και είμαι ανοιχτή σε προτάσει και προσθήκε. Επίση ευχαριστώ θερμά τη γραμματεία τη Επιτροπή μα για την υποστήριξη. Κρίμα γιατί κάποιε σημαντικέ μελέτε ήρθαν πολύ αργά. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Εύχομαι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να δείξουν την ίδια ανοιχτή στάση στην ε, έκθεση του Κοινοβουλίου και να υπάρξει συνεργασία. Η Κυπριακή Προεδρία, με την οποία είχα έτυπες επαφές, αναγνωρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου και θεωρεί ότι με κάποιες προσθήκες από τα αιτήματα του Συμβουλίου μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ακόμα και αντιπαράθεση, αν θέλει το καθένας ε, ε, έχει να πει τη δική του οπτική γωνία. Είναι δύσκολο να βρει ισορροπίε για τέτοια πρόταση. Όμω, εν τέλει, θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα πλειοψηφικό κείμενο που είναι ισχυρό, ώστε να μπορέσει να ισχυρή πρόταση τη Επιτροπή Πολιτισμού, ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε και το πρόγραμμα και το προπολογισμό του. Γιατί με τι ειδήσει που λαμβάνω τι τελευταίε μέρε, αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Καβαντά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Με πολύ προσοχή άκουσα την παρουσίαση της Σίλβια και θα ήθελα ειλικρινά να την ευχαριστήσω για την πολύ δύσκολη δουλειά την οποία έχει κάνει. Νομίζω ότι ε, προβλέπεται μία ακόμα συνάντηση σήμερα το βράδυ, δεν κάνω λάθος πολύπλοκο το ζήτημα αυτό γιατί προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδυάσει δύο διαφορετικά προγράμματα και από την άλλη κάνει και μία πρόταση κανονισμού. Με αποτέλεσμα νομοθέτης να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση καθότι πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πολύ γενικό, κατά την άποψή μου αόριστο κείμενο και σε πολλά σημεία συγκεχημένο. Έχω ενημερωθεί από την εισηγήτρια ότι έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και ότι προσπάθησε να πετύχει μια ισορροπημένη θέση. Είμαι σαφώς υπέρ του, της ισορροπίας που επιτυγχάνεται, υπέρ του προγράμματος πολιτισμός. Η στάση που είχε κρατήσει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν ε, λογική πιστεύω και ούτε ανταποκρινόταν στις απαιτήσει των εκπροσώπων του τομέα του πολιτισμού και του, του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία τα οποία παραμένουν συγκεχημένα. Δεν γίνονται, για παράδειγμα, συγκεκριμένε προτάσει όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο. Εφόσον πραγματικά μιλάμε για πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πρόταση κανονισμού, την οποία εξετάζουμε σήμερα, θα αποτελέσει την νομοθετική βάση για ένα μέσο το οποίο θα καθορίσει το μέλλον του πολιτιστικού και όπτικου ακουστικού τομέα για τα επτά επόμενα χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, πραγματικά θα βαδίσουμε σε πολύ άγνωστα εδάφη. Πιστεύω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε καλύτερα αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Χρειάζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο, επιβάλλονται συγκεκριμένε δράσεις προκειμένου να καταφέρουμε να διασκεδάσουμε όλες αυτές τις ασαφείς ζώνες που υφίστανται στην πρόταση. Πρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής πού πηγαίνουμε και θεωρώ ότι στο, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ξεκαθαρίζεται αυτό. Επίσης, βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η πρόταση κανονισμού πολλές φορές αόριστα και σαφώς αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά προγράμματα χωρίς να υπάρχει άμεση διασύνδεση μεταξύ τους. Γίνεται μία αναφορά σε τοπικά περιφερειακά προγράμματα, στην πληρωμή συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην υπεκπροσώπηση των γυναικών στον πολιτιστικό τομέα, στο συσχετισμό ανάμεσα στον πολιτισμό και την κατάρτιση στην εκπαίδευση και την πανεπιστημιακή παιδεία. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν βρίσκουν απαραίτητα όλα αυτά την κατάλληλη θέση στα πλαίσια ενός προγράμματος πλαισίου. Επίσης, χρησιμοποιούνται κάποιες έννοιες νέες, οι οποίες δεν είναι σαφείς. Πολλές φορές είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιες θα είναι οι δράσεις οι οποίες θα σχετιστούν με τις έννοιες αυτές. Ενεργό συμμετοχή, δημιουργική εταιρική σχέση, είναι μερικές από τις νέες έννοιες που χρησιμοποιούνται Επίσης, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε προσεκτική αναφορά στην συμμετοχή των τρίτων χωρών στα πλαίσια του προγράμματο Media. Και Σίλβια, θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω για ποιο λόγο εσεί, ε, στην τροπολογία σα 160 ε, έχετε διαγράψει τη σχετική αναφορά. Θα μιλήσουμε πάντω για αυτό σήμερα το βράδυ, φαντάζομαι. Θα ήθελα επίση να γνωρίζω επίσης και την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Για ποιο λόγο διαγράφει η αναφορά στην ε, τροπολογία 160. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν κάποια πολλά θετικά σημεία τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε. Είναι πολύ σημαντική είναι πολύ σημαντικός ο καταμερισμός στον προπολογισμό όπως προτείνεται από την εισηγήτρια, το ότι αποσαφηνίζεται ο καθεστώς το οποίο θα έχει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο στον οπτικοακουστικό τομέα και το γεγονός ότι γίνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια. Επίση θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν έχει αντιμετωπίσει σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραμένουν πάρα πολύ αόριστα. Η εισηγήτρια προσπάθησε να ε, επιφέρει κάποιες αλλαγές, να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Παρ' όλα αυτά δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το προτινόμενο σύστημα και το πρόγραμμα αυτό πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτό ακόμα βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από την βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος. Δεν ξέρω αν τελικά θα προωθήσουμε καλύτερα ένα πρόγραμμα πολιτισμού και ένα πρόγραμμα μέντια μέσω ενό συστήματος το οποίο θα παρέχει εγγύησει. Φοβάμαι ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς μια εμπορευματοποίηση αν θέλετε των τομέων αυτών. Μέσα από τις τροπολογίες μου θα δείτε τις παρατηρήσεις μου αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και πώς θα λειτουργήσουν στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε. Μας λέει σε πολλά σημεία ότι θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία και ότι θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις νομοθετικές πράξεις αλλά αυτό το οποίο λέω κάθε φορά για το ζήτημα αυτό, δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε σε καμία περίπτωση λευκή επιταγή για τα ζητήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ούτε σήμερα πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Σας ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Και επίση θεωρώ ότι δεν είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εφαρμόσει στον πολιτιστικό τομέα ένα χρηματοδοτικό μέσο όπως αυτό ακριβώς προβλέπεται για τις υπόλοιπες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγορές δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ένα χρηματοδοτικό μέσα το οποίο θα προβλέπει ένα σύστημα εγγύσεων μπορεί ενδεχομένως να είναι θετικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο συμφέρον και τόσο ενδιαφέρον τελικά για τους παράγοντες, ε, με συγχωρείτε, τους φορείς που ε, δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος ε, του τομέα του πολιτιστικού θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα στις διαφορετικές αγορές και θα πρέπει στον πολιτιστικό τομέα να έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε σωστά τον πολιτιστικό τομέα, όπως ακριβώς το κάνουμε και στον τομέα media. Α μην ξεχάσουμε ειδήσει στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε μπορεί ενδεχομένω να περιθωριοποιηθούν. Φανταστείτε, για παράδειγμα, πώ θα καταφέρει να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο ένα μικρό πολιτιστικό φορέα από μία μικρή πόλη, που ενδεχομένω όμω να έχει να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Κατά την άποψή μου δεν θα καταφέρει να έχει πρόσβαση. Επίση, το 11% που προβλέπεται στο Ταμείο Εγγύσεων και αυτό θεωρώ πάλι ότι μπορεί να μην λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για χρήματα, πιστώσει που δίνουν οι τράπεζε, απλώ αναφερόμαστε σε μια εγγύηση. Και στο νέο αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να ληφθεί ε, υπόψη όχι μόνο ο νέο προπολογισμό που θα προβλέπεται για τι ε, ευρωπαϊκέ ε, πολιτιστικέ πρωτεύουσε, αλλά και ένα νέο προπολογισμό που θα προβλέπεται για το νέο ευρωπαϊκό πολιτιστικό σήμα. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τις ε, νέες συμμετέχουσες χώρες και καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των διαφορετικών συνιστοσών μπορεί να οδηγήσει σε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Ενδεχομένως η πρόθεσή σας ήταν πολύ θετική, αλλά στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε κάποια σημαντική προστιθέμενη αξία. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι δεδομένη τη σημασία του κειμένου αυτού, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή στο κείμενο αυτό. Και αυτό ακριβώ τον ρόλο εμεί πρέπει να διδραματίσουμε ω συνομοθέτε. Προσπαθήσαμε αυτό να το κάνουμε και με άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε εξετάσει στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να διευκρινίσουμε όλες τις πτυχές της πρότασης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας καθοδηγήσει στη δουλειά την οποία θα κάνουμε. Τρεις ε, άξονες εργασίας έχω εγώ όσον αφορά την ε, σύνταξη των ε, τρυπολογιών. Πρώτον, να ξαναδώσουμε στην πρόταση αυτή έναν προσανατολισμό καλύτερο, πιο συγκεκριμένο και που θα περιέχει μια καλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο προγράμματα, πολιτισμός και μίντια και θα πρέπει για κάθε πρόγραμμα να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλει να κάνει η Ευρώπη για κάθε πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι ακόμα σαφές αυτό. Δεύτερον, να υιοθετήσουμε ακριβώς το πεδίο εφαρμογή του κάθε προγράμματος, διευκρινίζοντας ακριβώς τις μελλοντικέ δράσεις και δίνοντας συγκεκριμένου ορισμούς. Και τρίτος άξονας, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή του ε, εγκυοδοτικού προγράμματος χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών, να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε με έναν τρόπο συγκεκριμένο και πρακτικό, ρεαλιστικό, τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους ε, τομείς αυτούς. Θα μιλήσουμε λοιπόν και πάλι με την ε, Σίλβια, προσπαθώ να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και βέβαια θα σας βοηθήσω εγώ σε αυτό, να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Κύριε Συγήτρια, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Madame Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Σίλβια για την εργασία που έχει κάνει. Εξαιρετική πραγματικά εργασία για ένα κείμενο ιδιαίτερα πυκνό και πολύπλοκο. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε πρόταση είναι υπέρ της πρόθεσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι πρόσδεκτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση ως το δυνατόν περισσότερων Ευρωπαίων πολιτών και φορέων όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία υφίστανται ή δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα από την πιο νεαρή ηλικία δυνατόν. Συμφωνώ με τον κύριο Γκαβαντά ότι θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ πιο λεπτομεριακοί και συγκεκριμένοι όσον αφορά τα καλλιτεχνικά έργα, όσον αφορά την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τους καλλιτέχνες, την δυνατότητα να μπορούμε να προωθήσουμε τόσο το πρόγραμμα πολιτισμός όσο και το πρόγραμμα Μέντια. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την προώθηση νέων οικονομικών και πολιτιστικών μοντέλων, την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα καλλιτεχνικά έργα, καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην χρηματοδότηση όσον αφορά όλο τον καλλιτεχνικό τομέα, καλύτερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε την ε, διάχυση όλων των καλλιτεχνικών ε, πολιτιστικών έργων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όσον αφορά τώρα το δίκτυο στο οποίο αναφερθήκατε, νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε το δίκτυο αυτό και για τις διεπαγγελματικές επαφές και για τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέα διεθνικά σχέδια στον τομέα του πολιτισμού. Και επίση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα για τη δημιουργική Ευρώπη να συνάδει και με άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ευρώπης, κυρίως με την πολιτική συνοχή. Μέσω τη πολιτικής συνοχή προβλέπονται πολλές νέες δυνατότητε χρηματοδότησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά τώρα την την αξιολόγηση. Νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε πραγματικά στα χέρια μας ένα πρόγραμμα το οποίο θα προωθεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θα πρέπει να αποτελεί όμως και ένα πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία όσον αφορά το τομέα του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμούμε επίσης να έχουμε μια κάποια ευελιξία όσον αφορά τον επιμερισμό της εργασίας που θα πρέπει να γίνει, ιδίω αν συμπεριλάβουμε και νέους τομείς στο πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Μάρκος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί το έργο που μας παρουσίασε σήμερα η κυρία Κώστα είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά. Εδώ και ένα διάστημα το παρακολουθούμε ιδιαίτερα ε, στη χώρα μου, καθώς προσπαθούμε να καταστήσουμε κοινωνού στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου στο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, μια ε, κοινή πρόταση και ως ε, πολιτική ομάδα αλλά και ως κοινό συμφέρον. Όπω έλεγε πριν από λίγο ο συνάδελφο κ. Καβαντά, η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Δημιουργική Ευρώπη σίγουρα διαφέρει σημαντικά και από τον έρασμο για όλους. Γιατί αν στον έρασμο υπήρχαν κάποια σημεία που ως κοινοβούλιο, ως πολιτική ομάδα δεν ε, ασπαζόμασταν, παρά τα αυτά υπήρχε μία διάρθρωση και δομή σαφής. Σε ό,τι αφορά την δημιουργική Ευρώπη, αντιθέτως, φοβούμε υπάρχουν σκέλη αρκετά θολά και λιγότερο κατανοητά για πολλούς για το πώς θα μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Σκόπιμο λοιπόν είναι να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το φάκελο. Και πέρα από τη δουλειά που έχει γίνει έως σήμερα, πόσους ασχολήθηκαν με την πρόταση αυτή. Να δούμε βεβαίως και πώς θα πάει η συνάντηση ανάμεσα στην κυρία Κώστα, τον κύριο Καβαντά και τους λοιπούς σκιώδεις, θα είναι και όλοι οι άλλοι παρόντες. Ωραία. Οπότε Ας δούμε αν από αυτή τη συνάντηση που θα έχουν απόψε ξεπεραστούν τα μείζωνα προβλήματα. Οπότε να δούμε και εμείς ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή ε, Πολιτισμού θα προχωρήσουμε πριν δώσουμε σαφές χρονοδιάγραμμα. Ε, ε, Χάνω τάκουλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πολύ σύντομα δύο λόγια για την έκθεση της κυρίας Κώστα. Κάποιες δικές μου σκέψεις και κάποιες σκέψεις του Σκιώδους που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Λοιπόν, κάποιες προσωπικές δικές μου σκέψεις καταρχήν. Εδώ υπάρχουν τρεις θεματικές που αλληλοϊποστηρίζονται σε ένα ευέλικτο πλαίσιο. Πράγμα που αποτελεί πρόοδο στον οπτικοακουστικό τομέα. Υπάρχουν καινούργιες μορφές συνεργασίας. Αν πρέπει να οριοθετήσουμε μεταξύ πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα και μετά μεταξύ των οργανισμών που είναι εμπορικές ή όχι, ίσως αυτό να μην έχει και τόσο νόημα να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η ευελιξία που θα μπορούμε να έχουμε. Χρειάζεται ένα κοινό πρόγραμμα που θα μπορέσει να υποστηρίξει όλη αυτή την ποικιλομορφία του πολιτισμού, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, σύντομα κάποια επιμέρους. Ε, αναφέρομαι στις τροπολογίες για, τον, ε, την πολιτιστική ποικιλομορφία που υπάρχει στην 39-40 ε, τροπολογία. Είναι σημαντικό να τα στηρίξουμε αυτά. Πάντως πιστεύω ότι ο οπτικοακουστικός τομέας δεν πρέπει εδώ να αναφέρεται ξεχωριστά, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα στην 44 τροπολογία, εδώ μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα. Εγώ όμως περιορίζομαι σε μία ερώτηση. Υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ειδικά τις γυναίκες εδώ. Υπάρχει κάποιος λόγος ναι, οι άλλες ομάδες, ε, ε, άτομα με αναπηρίες, ναι, θα πρέπει να αναφερθούν στα προγράμματα αυτά. Άτομα με ειδικέ ανάγκες, λέει εδώ. Ε, κάποια ένωση ατόμων με ειδικέ ανάγκες ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου είπε ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα. Η ευελιξία, όπως προείπα, είναι σημαντικό πράγμα και επί της ουσίας πρέπει να πω ότι πάμε πράγματι εδώ στη, προς τη σωστή κατεύθυνση. Να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί σε όλα αυτά τα προγράμματα Εδώ διαφοροποιούμε λίγο σε σχέση με την εισηγήτρια, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία, αλλά οι δομές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να είναι μεγαλύτερα τα προγράμματα. Και είναι σημαντική η συνεργασία. Δεν θα πρέπει να βάζουμε όρια και να περιορίζουμε κάποιο πρόγραμμα επιμέρους. Αν όμως θέλουμε να είμαστε και αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, χρειαζόμαστε και περισσότερα χρήματα. Τα διάθετα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλά. Αν δεν διατεθούν σε ένα πρόγραμμα δηλαδή. Τέλος να τονίσουμε ότι το συνολικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες. σε ό,τι αφορά δηλαδή τα πολιτιστικά θέματα. Η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική για τη διάθεση των πληροφοριών. Οι μεταφράσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί έτσι μπορούμε να ε, μπούμε καλύτερα μέσα στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι και σε αυτό και σε άλλα θέματα συνεργάστηκα πολύ καλά με την κυρία Κώστα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα να πω και εγώ κάποια πράγματα. Το θέμα των γυναικών με ενόχλησε και εμένα λίγο, αναφέρομαι στην ε, τροπολογία 14. Δεν ξέρω, η Κομισιόν που προωθεί επιμέρους καλλιτέχνες. Ούτε εδώ προωθεί ε, καλλιτέχνες ε, άρενες ή γυναίκες. Η Κομισιόν προωθεί πολιτιστικά προγράμματα που εντάσσονται οι μεν και οι δε ή οι μεν ή οι δε. Γι' αυτό βεβαίω και οι γυναίκες να υποστηρίζονται στο βαθμό που είναι καλές. Αλλά δεν θέλω να φορτώσει το πρόγραμμα ε, με κάτι που δεν του ανήκει, δηλαδή δεν είναι δουλειά του. Έτσι αντιδρώ εγώ. Και νομίζω ότι και η αναφορά στους άτομα με αναπηρίες δεν κολλάει. Χρειάζεται προσοχή. Αυτό το πραγματικά μικρό πρόγραμμα που έχει δύο συγκεκριμένους προσανατολισμούς, από τη μια το σκέλος των πολιτιστικών προγραμμάτων και από την άλλη τα μέσα και το οπτικοακουστικά, ε, μην το φορτώνουμε υπερβολικά με πολλά μικρά πράγματα τα οποία βεβαίως είναι σημαντικά για την καθημερινή ζωή. Αλλά θα δυσχερανθεί το πρόγραμμα το ίδιο πρέπει να πω και για το δικό μου πρόγραμμα, ε, για το άλλο πρόγραμμα που έχω αναλάβει, που ε, έχω δεχθεί εκεί 500 τροπολογίες και δεν ξέρω τι να τις κάνω. Εν πάση περιπτώσει χρειάζονται βασικοί άξονες μεγάλοι, όπως είπε και ο κύριος Κάβαντα, θα πρέπει να δείχνουν άμεσα ε, πού προσανατολίζονται, τι εννοούν και τι πρέπει να καταλάβουμε. Αυτά είχα να πω εγώ και ρωτώ την Κομισιόν σε αυτό το σημείο. Ποιο θέλει να μιλήσει από την Κομισιόν, ο κύριο Δρούσα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαιρετίζει την έκθεση της κυρίας Κώστα στο βαθμό που υιοθετεί το γενικό πνεύμα για τη βασική αρχιτεκτονική της πρότασης της Κομισιόν, ενσωματώνοντας ε, όλη την υποστήριξη για τους ε, ε, καλλιτεχνικούς τομείς, τους οπτικοακουστικούς, προβλέποντας νέο δημοσιονομικό μέσο, διευκόλυνση και αυξάνοντας για τον προϋπολογισμό. Η έκθεση αλλά και η συζήτηση δείχνουν ότι μεγάλη προσοχή έχει δοθεί σε κάποια θέματα και προβληματισμούς που αποτέλεσαν τη βάση και της πρότασης της Κομισιόν. Η ανάγκη να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της ενδογενούς εσωτερικής αξίας του πολιτισμού και της συμβολής της στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να τονίσω ότι, για παράδειγμα, το μέσον που προτείνεται με αυτό το... Δεν είναι αντίγραφο πιστό του μέσου το οποίο ε, εφαρμόζεται στο πρόγραμμα Media. Είναι άλλο μέσο μεγαλύτερο σε πεδίο εφαρμογής με προσέγγιση χαρτοφυλακίων και με δυνατότητα ικανο... δημιουργίας οικοδόμησης ικανοτήτων επίσης. Και τη δοκιμασία στην αγορά που γίνεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων δείχνει ότι αυτό προχωρά πολύ τον οπτικοακουστικό τομέα και τον ε, τομέα που είναι εμπορικό. Πρέπει επίσης ε, να ληφθούν απόλυτα υπόψη οι ιδιαιτερότητε του τομέα του πολιτισμού αφενός και του οπτικοακουστικού από την άλλη. Η Κομισιόν δεν ζητάει λευκές επιταγές και μάλιστα αν δείτε την πρόταση και συγκρίνετε το τωρινό, το, τους στόχους του πολιτιστικού προγράμματος του τωρινού και την ε, δημιουργία για την Ευρώπη βλέπουμε Τη δημιουργική Ευρώπη βλέπουμε ότι τα κριτήρια για το πολιτιστικό σκέλος είναι πολύ πιο λεπτομερή και εξειδικευμένα από ό,τι στο τωρινό πολιτιστικό πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να βρούμε ευκαιρίες για να διευκρινίσουμε τις συστάσεις, αλλά η πρόκληση εδώ νομίζω ότι θα είναι να υπάρξει ισορροπία αποφεύγοντας ε, έναν αριθμό κινδύνων. Ο πρώτος κίνδυνος, και νομίζω κυρία Πρόεδρε τον αναφέρατε λέγοντας ότι δεν πρέπει να παραφορτώνσουμε το πρόγραμμα αυτό, και πράγματι πρέπει να φροντίσουμε να μην επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του πέρα από αυτά που μπορεί να παραδώσει, πέρα από τα παραδοτέα του αν θέλετε. Και εδώ έχουμε κάποιες ερωτήσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος εις ό,τι αφορά τον τομέα, αναφέρει τον τομέα της μόδας. Εμείς καλύψαμε το κομμάτι του σχεδιασμού, design, στην τωρινή μας πρόταση, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι πρέπει να καλύψουμε και όλη τη μόδα. Εις ό,τι αφορά τους στόχους και τις δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές έννοιες που είναι ευρύτερες από τους στόχους του προγράμματος. Υπάρχουν αναφορές σε εκπαίδευση, κατάρτιση, πανεπιστήμια σε πολλά σημεία και ίσως αυτό δεν είναι το καλύτερο πρόγραμμα για να τα πούμε όλα αυτά. Επίσης μιλάμε για τον ε, ψηφιακό γραμματισμό που χρησιμοποιείται και που είναι πολύ ευρύτερος από ότι το γραμματισμό των μέσων γίνεται αναφορές στις τοπικές εξελίξεις, στην διασυνοριακή διαεθνική ε, συνεργασία που ξεπερνά επίσης το πρόγραμμα. Επίσης μιλάμε για υποστήριξη των ε, καλλιτεχνικών εκφράσεων, πολιτιστικών εκφράσεων και την διαφύλαξη της κληρονομιάς μας. Δεν νομίζω όλα αυτά μπορεί να τα καταφέρει το πρόγραμμα. Ο, στη διατύπωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτω ώστε να μην το παραφορτώσουμε όπως είπαμε. Ένας άλλος κίνδυνος είναι... Ε, να αποφύγουμε ε, ε, ε, τα προβλήματα υλοποίηση. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Μιλήσατε για την προτεραιότητα στι γυναίκε. Αυτό και για την υλοποίηση θα ήταν προβληματικό για ένα πρόγραμμα που στηρίζει οργανισμούς και όχι άτομα. Επίσης, κάποια πράγματα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα με δείκτες, θα έχουμε τα δεδομένα. Θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα παραφορτώσουμε με πολύ μικρούς οργανισμούς με αυτή την υποχρέωση να μας δίνουν τα δεδομένα. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται προσοχή τι δεδομένα ζητάμε. Ο τρίτος κίνδυνος που θέλουμε να αναδείξουμε είναι ο κίνδυνος της, ε, των δισκαμψιών, των ακαμψιών. Όπως είπαμε, μιλάμε για πρόγραμμα που θα έχει επταετή διάρκεια μεσούσης της κρίσης και των αλλαγών. Και δεν είμαστε βέβαιοι, για παράδειγμα, ε, αν βάλουμε ανώτατο όριο στο 75% που δεν ε, συνάδει με την τρέχουσα πρακτική στο πρόγραμμα ε, πολιτισμός και μέσα, ε, δεν ξέρω αν είναι καλή πρόταση. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι γιατί οι προϋπολογισμοί των πολιτιστικών οργανισμών ε, έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Το ίδιο αφορά και τις ε, τροπολογίες που αφορούν το παρατηρητήριο. Δεν, περιμένουμε, δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2015 για να ελέγξουμε αν υπάρχει διάθεση να διευρυνθεί η εντολή του παρατηρητηρίου. Και εδώ χρειάζεται ευελιξία λοιπόν. Ε, μια άλλη παρατήρηση τώρα. Η Κομισιόν δεν συμμερίζεται κατά πάσα πιθανότητα τη νομική ανάλυση του Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση του ετησίου προγράμματος εργασίας. Η Κομισιόν έχει αναλύσει το πρόγραμμα εργασίας, το περιεχόμενο ε, καθορίζεται από κανονισμούς και εδώ χρειάζεται εκτελεστική και όχι ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Και αυτή είναι η μόνη εκτελεστική πράξη που προβλέπει η Κομισιόν για να εφαρμοστεί η δημιουργική Ευρώπη. Ε, τέλος, να εκφράσω την προθυμία μας να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και για να αναπτύξουμε επικοδομητικές λύσεις όπου αυτές θα χρειάζονται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ξαναγυρίζω στο τελευταίο θέμα της κατε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Έχουν οριζόντια σημασία. Θα τις βρείτε σε κάθε πρόγραμμα. Εμείς κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε σε όλα τα άλλα προγράμματα. Δεν... Ε, ε, είστε βέβαια εσείς ο μόνος υπέρμαχος, έχετε και, ε, και άλλους συνοδοιπόρους, όπως άλλωστε έχουμε και εμείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά θα γνωρίζετε ότι έχουμε εκλογέ στην Καταλωνία. Και σήμερα είχα κάτι δουλίτσες να τελειώσω στη Βαρκελόνη. Ήθελα να ακούσω και τον συνάδελφο Μπενέν Βάγε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν εδώ. Αλλά ξέρετε, αυτό το Σαββατοκύριακο ο κύριος Αμπέρ ήταν και γραμματέα αυτή τη επιστροφή και τώρα είναι επικεφαλή του γραφείου του Κοινοβουλίου στη Μαδρίτη. Αυτό ο κύριο λοιπόν έκανε μη, διοργάνωσε μια συζήτηση με 100 προσωπικότητε του πολιτισμού και τη τέχνη για να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και ήθελα να σα αναφέρω εντάχει κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν. Έτσι, εξ αρχή δεν άρεσε η ιδέα τη συγχώνευση προγραμμάτων. Δηλαδή, όταν το πρόγραμμα Κούλτ και το πρόγραμμα Μέντιελ λειτουργούν καλά, γιατί να συγχωνευτούν. Έπειτα, να γίνει αποδεχτό το κοινό πρόγραμμα, αρκεί να μιλήσουμε για τα διαφοροποιημένα προγράμματα. Έπειτα, ε, οικονομικές εγγύσεις είναι μια καλή ιδέα. Αυτό που δεν είναι σαφές και θέλω και εγώ να ρωτήσω κάποιες διευκρινήσεις, πώς θα δοθούν αυτές οι εγγύησεις, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Έπειτα, όλοι ρώτησαν κατά πόσον τα γραφεία που υπάρχουν σήμερα σε περιφερειακό επίπεδο θα διτηρηθούν, ώστε να παραποιημένει αποκεντροποιημένο το πρόγραμμα ε, Media και Cult. Γιατί πραγματικά θα είναι μία απώλεια αν το χάσουμε αυτό. Προσοχή λοιπόν, ε, προσοχή για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ που προσπάθεια noch was eingefallen, bevor ich Ναι, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα, θέλω να πω το εξή. Δεν καταλαβαίνω αυτό το λογότυπο των ε, μέσων, γιατί δεν θέλει η Κομισιόν να το χρησιμοποιήσει. Έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ταινίες που βραβεύτηκαν στηρίχθηκαν, υποστηρίχθηκαν από το Μέντια και Παντού υπάρχει αυτό ο λογότυπος που είναι μικρός και ωραίος. Και πρέπει τώρα να τον εξαφανίσουμε και να βάλουμε κάτι άλλο ή τι. Αυτό είναι αστείο. Δεν μου είχε απαντήσει κανείς. Η κυρία Σίλβα κουνάει το κεφάλι, άλλοι ε, κάνουν άλλες ε, χειρονομίες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Α, είναι, είναι κουτό να εγκαταλείψουμε κάτι που λειτουργεί ένα ωραίο λογοτυπάκι το οποίο ήταν γνωστό σε όλο τον κινηματογραφικό κόσμο. Να το, να το αφήσουμε, να το εγκαταλείψουμε γιατί. Για πείτε μου, εξηγήστε το μου αυτό εν συντομία. Βλέπω κάποιοι κυρίοι, παρακαθήμενοι σας κουνούσε το κεφάλι. Ε, πείτε μας, τι έχετε να μας πείτε πάνω στο λογότυπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για το λογότυπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, αποφάσισε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι οι πολίτες να βλέπουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ο πολλαπλασιασμός λογοτύπων στα κοινωτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θόλωνε την εικόνα. Και γι' αυτό αποφασίστηκε να ε, γυρίσουμε πίσω σε πολύ απλά λογότυπα που θα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σημαία. Τώρα για το πρόγραμμα Media, βλέποντας αν θέλετε την εμπορική αξία του λογότυπου, είπαμε, αποφασίσαμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος θα υπάρξει μια εξαίρεση που θα επιτρέπει τη χρήση αυτού του λογοτύπου. Για το μέλλον η πρόταση της Κομισιόν είναι εξακολουθεί να είναι για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίζεται η ανακοίνωση σε ένα λογότυπο με την σημαία της Ένωσης και την αναφορά του ονόματος του προγράμματος. Ελπίζω να σας ε, ε ξεκαθάρισα την άποψη της Κομισιόν εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Το Μέντια δεν είναι πρόγραμμα η κυρία, που, που το ξέρει η κυρία Ντυπών και η κυρία Πακ και η κυρία Τάδε και η κυρία Δίνα αφορά τον κινηματογραφικό κόσμο, τον κόσμο του κινηματογράφου, αυτούς που δουλεύουν καλλιτεχνικά σε αυτό το τομέα και όταν προβάλλεται η ταινία πάντα είχε το λογότυπο. Ποιον πείραξε, ε, δεν πειράζει να βάλουμε και το λογότυπο με τα στεράκια, αλλά αυτά που έχουν καταξιωθεί δεν χρειάζεται να τα πετάμε ξαφνικά ή να ε, τα βάζουμε όλα κάτω από τον ίδιο μανδύα. Δεν βοηθάει αυτό πρέπει να πω εκπείρασε. Εσείς ε, βέβαια μας ε, τα εξηγήσατε, απαντώ κι εγώ. Αλλά όποιο δεν δείχνει το μέντια με το πραγματικό του όνομα και το λογότυπό του, δεν έχει καταλάβει πόσο καλό ήταν το μέντια. Τώρα, η Σίλβια Κώστα. Βεβαίως ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια, ακόμα και για την ειλικρίνεια στα λόγια σας που ζητήσατε μεγαλύτερη σαφήνεια και διευκρινήσεις. Είναι απόφευκτο. Είναι απόφευκτο, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ για αυτή την κατανόηση. Ε, το θέμα είναι περίπλοκο και κανθώδες. Και είναι μια πρόταση που σε σχέση με άλλες φέρει μια πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με άλλα προγράμματα που είχαμε παραδοσιακά συνηθίσει έτσι. Αυτή είναι η ζωή και είναι αυτό κατανοητό. Από εκεί πέρα είπα ότι ανοιχτή και για αλλαγές και προσθήκες, ελπίζοντας να υπάρχει συμφωνία επί νέων προτάσεων που θα βελτιώσουν την έκθεση. Αυτό είναι λογικό με στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου. Όμως θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τη γενική προσέγγιση που αν καταλαβα καλά αυτό το ασπάζεστε, που είναι δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα στο να έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο, ο είπε ο κ. Καβεντά και η Σταθροπός επίσης, και είναι η καινοτομία εν προκειμένου καθώς περιέχει πραγματικά καινοτόμα στοιχεία σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα τη προηγούμενη αυταετία, αλλά λοιπόν, πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζοντα την αυτονομία των δύο προγραμμάτων, για να το πω και στον ε, κύριο Φίσο που ήρθε καθυστερημένο ότι ακριβώς αυτό κάνουμε. Δηλαδή, έτσι έχουμε χωριστά προγράμματα, χωριστούς δικαιούχους, χωριστή χρηματοδότηση και μέτρα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες, να το κάνουμε. Αλλά να διατηρήσουμε ένα επαρκές επίπεδο ευελιξίας. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κανονισμό που θα ρυθμίσει ένα τομέα που είναι σε μια διαδικασία δυναμικής αλλαγής. Τώρα, σε σχέση με κάποιε ανησυχίε που ακούστηκαν για κάποια επιμέρου σημεία, σε ό,τι αφορά κάποιε επιμέρου διατυπώσεις, εκφράσει που κατά την κρίση είναι πολύ κοινέ φράσει, κοινή γλώσσα στα ευρωπαϊκά έγγραφα, αλλά και σε θέματα πολιτισμού, αλλά και νέε έννοιε που εμφανίζονται. Π.χ. Αυτό που επέλεξα τι για audience building στα αγγλικά, να μιλήσουμε για audience development πάντοτε στα αγγλικά, βασίζεται σε έναν προβληματισμό που ακριβώς βασίζεται στον τρόπο τον οποίο προάγουμε πλέον τον πολιτισμό και δεν έχουμε να κάνουμε με τη δημιουργία μιας αγοράς, δημιουργία ενός audience, ενός ακροατηρίου, αλλά και το άνοιγμα σε νέους ε, στόχους, σε, νέα ακροατήρια στόχους δεν είναι κάτι έτσι γενικό και αόριστο. Αντικατοπίστε κάτι συγκεκριμένο. Έπειτα, οι συμπράξει που προσπάθησα να εξηγήσω και πριν, οι δημιουργικέ συμπράξει. εξηγούσα και πριν ότι έχουμε να κάνουμε περισσότερους φορεί κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θέλουν να συμμετάσχουν σε μια σύμπραξη. Σκεφτείτε παράδειγμα τα μουσεία. Μια δημιουργική σύμπραξη τι σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο έναν νέο φορέα μίας φύσεως, αλλά και διατομιακά περισσότεροι από ένας φορέας μπορούν να προάγουν ένα νέο project. Και στο τοπικό επίπεδο, ο κ. Καβαντά είπε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω το εξή. Ξέρω πολύ καλά τι ανήκει και είναι αρμοδιότητα των ιδρυτικών Ταμείων και έχετε δίκιο, έχετε δίκιο και τι ανήκει στο Ταμείο συνοχή, ακριβώ γιατί μιλάμε και για ένα άλλο όγκο κονδυλίων, έτσι. Αλλά κάποια προγράμματα που ενώ μεν είναι καθολικά και αγκαλιάζουν τα πάντα, ταυτόχρονα έχουν και μια ε, πολύ σαφή τοπική συνιστόσα. Σκεφτείτε συγκεκριμένε πολιτιστικέ πρωτοβουλίε. Κάτι που ξεκινά τοπικά και ε, σιγά σιγά κερδίζει έδαφο πανευρωπαϊκά και αποκτά πανευρωπαϊκή διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν αυτό όταν ξεκινά τοπικά να χρηματοδοτηθεί από τα διευθυντικά ταμεία. Ξέρετε, είναι από τα πράγματα που το και περισσότερο ε, μέσα στα πλαίσια των νέων δημοσιομικών προοπτικών είναι ότι με αυτό το 1,8 δισεκατομμύρια που σίγουρα δεν αρκούν για αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διάδραση με τα κονδύλια που μπαίνουν στο Ταμείο Συνοχή, στα Ευκαταμία κτλ. Σκεφτείτε, αυτό που είπαν οι Επίτροποι Βασιλείου και Ταγιάννη που έκανε μια ανακοίνωση για τον κινηματογράφο και είπαν ότι θα ε, είναι πιο αλληλοσυμπληρούμενα τα κονδύλια τα οπτικοστικά μέσα με, και συμπληρωματικότητα με το Ταμείο Κόσμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια επικοινωνία, θα είναι πιο συγκοινωνούντα δοχή αν θέλετε πλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Φαίνεται ότι οι γυναίκες προκαλούν σκάνδαλο πάντοτε. Κοιτάξτε. Αν τώρα διατυπώθηκε στο κείμενο με τρόπο α, α, μη ε, α, σαφή, εγώ να το ξεκαθαρίσω όσο μπορώ. Απλά θέλω να πω ότι δεν μιλάμε επί πρόσθετες δράσεις, δεν ζητούμε πρόσθετε δράσει. Και πρόεδρε, έχετε δίκιο. Δεν εννοούμε αυτό. Δεν κάνουμε ένα apartheid υπέρ των γυναικών. Απλά να λάβουμε υπόψη το εξή στοιχείο. Ξέρετε ότι όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να έχουν ω ρήτρα το gender mainstreaming. Δηλαδή να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη διάσταση του φύλου και να υπάρχει ευθυγράμμιση. Έτσι να προβλέπεται ένας τρόπος ε, μιας κάπως ισότιμης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Στην Ευρώπη 40% των ε, συνθετών μουσικής είναι γυναίκες. Στα ραδιόφωνα, στις ορχήστρες, ε, στις συναυλίες εκπροσωπούνται από το 0,5%. Ε, δεν μιλάω λοιπόν για συγκεκριμένη δράση, απλά να λάβουμε υπόψη σε τέτοιου είδους project, να δίνετε μια ιδιαίτερη προσοχή και στην ε, συμμετοχή, συμπαρουσία, όπως θέλετε πείτε, και στις γυναίκες. έναν τρόπο. Αν θέλετε, αν μπορείτε να μου προτείνετε μια άλλη διατύπωση, βεβαίω να το κάνουμε. Δεν μιλάμε για άλλη δράση. Τώρα κάτι άλλο που ακούστηκε εκπαίδευση, πανεπιστήμια κτλ. Ευχαριστώ θερμά ε, τη συνάδελφο την κυρία Σάντζα Σμιτ για τις παρατηρήσεις της. Όσα είπατε. Ναι, ναι, θα μπορούσαμε να δώσουμε καλύτερη έμφαση ίσως ε, στο κείμενό μου, αλλά ήδη περιέχονται στο κείμενο όσα είπατε. Και βεβαίω έχετε και θέμενε απόψει. Ο ένα λέει ότι θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση στον τομέα τη ε, παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση. Ένα άλλο λένε όχι, δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Η Κομισιόν αυτό είπε τώρα. Ε, και εγώ πρέπει να βρω μια ισορροπία. Προσπαθώντα δηλαδή να κρατήσω την ευρωπαϊκή διάσταση της επαγγελματική κατάρτιση με τις ανταλλαγές, ε, τι μαθητείε κτλ. Και από την άλλη να μην ξεχάσουμε ε, την τον εγγραμματισμό μέσω των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη αν δεν υπάρχει καλύτερη καλλιέργεια του κοινού. Και εδώ το έχουμε ξαναπεί. Δεν είχαμε ξαναπεί να υπάρχει υποχρεωτικά στα σχολεία το φιλμ λιτέραση, κινηματογραφικός ε, γραμματισμός. Ε, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό εν προκειμένου σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να μπει και αυτή η διάσταση σχολεία. Δεν λέω όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο, σίγουρα. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκούρια για την κατανόηση που απέδειξε τα λεγόμενά του και θα μιλήσω και για τις προπτικές μετά. Για τον κύριο Τάκουλα. Α, με συγχωρείτε. Για τον κύριο Καβαντά, δεν ολοκλήρωσα. Να πω κάτι ακόμα. Φυσικά και θέλω πάρα πολύ να ξεκαθαρίσω κάποια α, κάποιες φαιές ζώνες, αν θέλετε, εδώ στο κείμενο. Βεβαίως, ό,τι είναι α, ασαφές θα πρέπει να διευκρινίσουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο κείμενο και μιλάμε εν προκειμένου για ένα κανονισμό. Και εφόσον μιλάμε για ένα κανονισμό που θα έχει διάρκεια ζωή σε 7 χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφή καθορισμό σε, σε επίπεδο στόχων, σε επίπεδο κονδυλίων στο τι ανήκει στο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, στα επιμέρους δύο υποπρογράμματα και τις πράξεις καταξιοδότηση. Και βεβαίως υπάρχει και ενδιάμεση αξιολόγηση στα μέσα του δρόμου. Πιστεύω αυτή είναι μια λογική δομή. Βεβαίω μπορεί να υπάρχουν και ε, διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει και αντίλογο. δεν ξέρω. Σήμερα με τους σκιώδε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και μπορούμε να βρούμε κάποιο κοινό έδαφος, πιστεύω. Για τον κύριο Τάκουλα, πολύ ορθά είπατε ότι θα πρέπει να βρεθεί μία μέση οδός ανάμεσα στα οπτικοακουστικά μέσα και τις άλλες πτυχές της πρότασης και σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ερωτήσεις που, ακού, ε, που ακούστηκαν, νομίζω ότι απάντησε ήδη η Πρόεδρος για τις πράξεις του Ουσιαδότης και συμφωνώ για την μόδα. Αν θεωρείτε ότι το design, ο σχεδιασμός καλύπτει την μόδα, Κάνετε όμως εσείς μια διάκριση ανάμεσα στην βιομηχανία και την δημιουργική παραγωγή. Ναι, αλλά η μόδα δεν είναι μόνο η βιομηχανία και η εμπορική πτυχή του πράγματος. Θυμηθείτε αυτό που έλεγε η Πράσινη Βίβλος ε, για την δημιουργία και την πολιτική δημιουργία. Ε, εγώ είχα την εντύπωση λοιπόν ότι η μόδα, επειδή είναι κομμάτι της δημιουργικότητας και του πολιτισμού, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Τώρα, για τη συγχρηματοδότηση. Τα προγράμματα που τρέχουν σήμερα προβλέπουν για κάποια ευελιξία. Δηλαδή, Συνήθω ο τελετή ε, συγχρηματοδότηση είναι 50% και μπορεί να ανέβει όμω στο 75% αν υπάρχει σαφή τεκμηρίωση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ευελιξία και πάλι. ευελιξία σε έναν βαθμό για να υπάρχει όμως και μία ομοιόμορφη προσέγγιση στα project. Για τα πανεπιστήμια να πω ότι μόνο μία φορά μνημονεύονται ως ε, μέσα του πολιτισμού, ε, φορείς πολιτισμού, ε, με τους οποίους μπορούμε να έχουμε συνεργασία σε προσπάθειες αλφαβητισμού, αγωγής του πολίτη κτλ. Πέρα από τις σχολές κινηματογράφου και άλλες επαγγελματικέ σχολές, από τα πανεπιστήμια, έχουν δημιουργήσει κάποια δίκτυα για όσους ασχολούνται με το κινηματογράφο. Και έλεγα ότι θα μπορούσαν να είναι και αυτοί εταίροι σε κάποια project. Αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερα. Δεν μιλούσα για μαθήματα στα πανεπιστήμια. Απλά να διευκρινίσουμε τώρα για το, την διεθνική συνεργασία και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Δεν καταλάβω την ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό ήδη θα πρέπει να προβλέπετε. Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε μια συνεργασία διαπεριφερειακή και διεθνική. Νομίζω ότι αυτό είναι και εκτιμένο δεδομένο. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σα. Σε ό,τι αφορά τώρα μια άλλη ερώτηση, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση φόβο που εκφράζατε, συνάδελφε, είπατε γιατί θέλετε να μειωθεί η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ή μάλλον ε, γιατί να μειωθεί η μαλλον γιατι τρίτων συμμετοχη τριτων φορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρόγραμμα Media, τη σχέση με την 160. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, το αντίθετο λέμε. Σήμερα τι προβλέπετε, να συμμετέχουν αυτές οι χώρες που ανέφερα πριν, και έπειτα με βάση διμερεί συμφωνίες μπορούν να προβλέπετε και συμμετοχή τρίτων χωρών με επιπρόσθετα κονδύλια και μέσω της πολιτικής γειτονίας μέσω συμφωνιών που ήδη υπάρχουν αυτές τις χώρες. Και είπαμε λοιπόν να διευρύνουμε, όχι να διευρύνουμε τον αριθμό των χωρών, να διευρύνουμε τους δικαιούχους. Να υπάρχει μια βαθμιαία προσέγγιση στην προσβασιμότητα. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Κάποιες χώρες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας οδηγής του 2010 χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια. Η Ελβετία χρειάστηκε πέντε χρόνια για να προσαρμοστεί από την πρώτη σταθερή οδηγία και αν κατάλαβα καλά, το ίδιο συμβαίνει και με την Κροατία. Άρα, έτσι, μεταξύ μας να το συζητούμε εντελώ φιλικά, σκόπι μου θεωρούμε θα ήταν για να μπορούμε να εγγυηθούμε την συνέχεια στην συμμετοχή αυτών των χωρών στο Μέντια να συμμετάσχουν και οι χώρες που είναι σχεδόν έτοιμες και όχι όσες ε, πληρούν όλους τους όρους. Ώστε να αποφύγει το εξή ε, γεγονός. Εκεί που θέλουμε να διευρύνουμε τη συμμετοχή αυτών των χωρών και σε αυτούς τους τομείς, ε, να θέτουμε όρους που καθιστούν αδύνατη τελικά την συμμετοχή τους. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σωστά διατυπωμένο αυτό, ότι σίγουρα κάποιες αρχές θα πρέπει πάντα να τηρούνται, εννοείται, αλλά αν θέλετε να το διατυπώσουμε. Αυτό ήταν το νόημα των λεγόμενων μου, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Εγγύησης. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι ένα οριζόντιο μέσο για πολλά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Είναι πολλά. Το Εράσμος, η Δημιουργική Ευρώπη, το Κόσμε κτλ όλα αυτά τα προγράμματα προβλέπουν να υπάρχονται σε αυτό α, εργαλείο εγγύησης. Όλα αυτά όμως έχουν δρομολογηθεί και είναι εξέλιξη. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ακόμα ε, τα επεξεργάζεται το Συμβούλιο, τα ακούει όλα αυτά τα στοιχεία η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο δεν έχει αποφασίσει και λέμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, λέμε τι είδους δάνεια και τα κονδύλια που δεν θα απορροφώνται θα επιστρέφουν στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Όλα αυτά τα λέμε στην έκθεσή μας και ανέφερα πριν και τους ενδιάμεσους, τους ε, χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους. Και αν μου λέτε αυτή είναι η τελική εικόνα, όχι, όχι, γιατί τους επόμενους μήνες το επόμενο διάστημα με αυτές τις ερωτήσεις που φτάνουν στην Κομισιόν και με τις προτάσεις που επεξεργάζει το Συμβούλιο, θα έχουμε πρόστα στοιχεία στη γενική εικόνα. Εγώ προσπάθησα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα στο μέτρο του δυνατού με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Αν θέλετε να βάλουμε και άλλε μεσαυτικές ρήτρε, να τι βάλουμε. Επειδή όμω μιλάμε για ένα χρηματοδοτικό μέσα, μέσο καινούριο, ή έχει πιλωτικό χαρακτήρα, το μέτιο που ξεκίνησε το 2009, αν θυμάστε, και λειτουργήσε για ένα χρόνο, Είχαμε δει ποια ήταν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και έγιναν πολλέ αλλαγέ. Προσπάθησα λοιπόν να κατανοήσω αυτή την αναγκαιότητα που γεννήθηκε το 2009, να διευκρινίσουμε δηλαδή κατά πόσον είναι χρήσιμο και υπό ποιου όρου. Είναι όμω μια ευκαιρία πιστεύω. Και πολλοί ενδιαφερομένοι φορεί βλέπουν αυτό το χρηματοδοτικό μέσο ω μια ευκαιρία Αυτή η διευκόλυνση λοιπόν που παρέχει αυτό το χρηματοδοτικό μέσο που λειτουργεί ως εγγύηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δοθεί μια όθηση σε αυτούς που χρειάζονται ε, μια τέτοια όθηση για να μπουν στην αγορά θα περιμένουμε να δούμε και την διάμεση αξιολόγηση βεβαίω για να δούμε κατά πόσον όλα αυτά που ε, αναμένουμε θα γίνουν πραγματικότητα. Προσπάθησα να τηρήσω και του χρόνου, λέει μιλήτρια. Αυτά από μένα. Είμαι στη διάθεσή σα. Απόψε έχουμε μια συνάντηση με τους Shadows, με τους Σκιώδης. Να πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ είμαι ανοιχτή να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ελπίζω όμως αυτό να μην πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ Σίλβια. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαβουλεύσεις από ό,τι φαίνεται ακόμα. Προτείνω 23 Οκτωβρίου να είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών όπως προτείνεται και να ψηφίσουμε το Δεκέμβρη. και τη δική μου έκθεση Yes Europe την αναβάλαμε. Γιατί κάνουμε προγράμματα επταετή. Πρέπει λοιπόν να μην βιαζόμαστε. Να πω κάτι ακόμα. Μην παραφορτώνουμε τα προγράμματα με πράγματα που δεν τα αφορούν και δεν έχουν σχέση με τα προγράμματα. Και ο αναλφαβητισμός και ο αναλφαβητισμός των μέσων δεν έχει να κάνει με εκπαίδευση κατάρτιση θα πάει στο πρόγραμμα Yes Europe. Το Media και ο πολιτισμός δεν είναι σχετικά προγράμματα. Ή η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ταιριάζει στο Εράσμου, στο Yes Europe. Καταλάβετε το παρακαλώ. Τα λίγα λεφτά που έχουμε είναι για ένα μικρό πρόγραμμα. Αν το παραφορτώσουμε αυτό το μικρό πρόγραμμα με όλα αυτά που μας είναι προσφυλή, αλλά που όμως δεν συγκαταλέγονται εκεί, αλλά συγκαταλέγονται για παράδειγμα στο Yes Europe πρόγραμμα, ε, τι να κάνουμε, πρέπει αυτά να τα λέμε όλα, αλλά να ξέρουμε ότι θα πάνε σε άλλα προγράμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά των γυναικών ή ότι δεν ε, θέλουμε τον ψηφιακό γραμματισμό αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ο κόσμος σε αυτούς τους τομείς με αυτό το πρόγραμμα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ε, εδώ συμφωνώ με την Κομισιόν. Δεν μου συμβαίνει και συχνά, δεν συμφωνώ μαζί της τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά πάντως χρειάζεται εδώ προσοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες που το, σκέφτηκαν πολύ το θέμα αυτό. Τις επόμενες 8 μέρες να συνεργαστούν καλά, να εξετάσουν και τις ε, ιδέες του κυρίου Καβαντά, να τις λάβουν υπόψη. Καλό είναι να βρεθεί κάποια συνένεση εδώ και παρακαλώ όλους τους συνεργάτες των ε, κυρίων και κυριών να ε, παρακολουθούν το θέμα και να δουλέψουν προς την κατεύθυνση συμβιβαστική λύσης για να μην κάνουμε αέναες συζητήσεις πριν από τις ψηφοφορίες και να έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα. Έτσι πρέπει δηλαδή να Συμπλέψουν οι απόψεις. Ωραία, καλή επιτυχία. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ πρόκειται για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Ξέρετε όλοι αγαπητοί μου συνάδελφοι ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα με μεγάλο αποτύπωμα. Είχαμε τη συζήτηση ότι δηλαδή αυτό δεν είναι πρόγραμμα για να το σχολιάσουμε, αλλά είναι ένα πρόγραμμα όπου θα πρέπει να πούμε ναι σε μια πρόταση ε, της Κομισιόν ε, του Συμβουλίου, διαδικασία έγκρισης. Ε, δεν γίνεται όμως και έτσι μόνο, άρα το εξετάσαμε. Το εξετάσαμε και η Νομική Επιτροπή και η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας είπαν μόνο σήμαντα ότι πρέπει να ισχύσει η συναπόφαση και όχι η έγκριση και το ανακοινώσαμε στην Κομισιόν ότι εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα και ορίσαμε και εισηγητή ο οποίος έχει υποβάλει έγγραφο στα πλαίσια όμως της συναπόφασης. Και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Τάκουλα για να μας πει τα σημαντικότερα πράγματα που θέλει να αλλάξει. Ε, μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να κάνουμε και συζήτηση αρκετή. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη για τους πολίτες είναι από τα σημαντικότερα προγράμματα. Αν και ο προϋπολογισμός του δεν είναι πολύ, 229 εκατομμύρια έχουν διατεθεί και πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα ήταν σημαντικό για τους πολίτες. Τολμώ να πω ότι έδωσε και προστιθέμενη αξία και όλοι γνωρίζουμε ε, ότι προσπαθούμε να τονίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, την αίσθηση της ιστορίας, την κατανόηση της ιστορίας, της ε, αδελφοποίησης πόλεων και αυτά χρηματοδοτούνται από αυτό το πρόγραμμα, από αυτό το πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ε, ότι αυτό είναι το μοναδικό πρόγραμμα όπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θέλουμε να προωθήσουμε ακριβώς αυτά τα πράγματα που σας είπα. Και η πρόταση αυτή είναι παρόμοια όπως το πρόγραμμα που τρέχει τώρα. Και πριν από πέντε χρόνια πάλι ήμουν εισηγητής γι' αυτό. Όπως ανέφερε η κυρία Πρόεδρος, είχαμε κάποιους διαπληκτισμούς και διαφορές σχετικά με το πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Πάντως, τώρα ε, στηρίχθηκε στη διαδικασία της συναπόφασης και ελπίζω και πιστεύω ότι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ομονοήσουν και ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν με τρόπο ευέλικτο. Θέλω να τονίσω ακόμη ότι η πρόταση αυτή είναι αρκετά καλή πέρα από το θέμα της νομικής βάσης και το Συμβούλιο έχει υποβάλει και καλές ε, τροπολογίες. Θέλουμε βέβαια να τεθεί έγκαιρα σε εφαρμογή το πρόγραμμα και εγώ εξέτασα και το κείμενο του Συμβουλίου το καλοκαίρι το στείλαμε και στους κοιόδης εισηγητές. Η έκθεση δηλαδή τώρα του Συμβουλίου υπάρχει σε όλες τις γλώσσες και μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση και να τη διαβάσετε. Οι δικές μου τροπολογίες αφορούν κάποια σημαντικά θέματα όπως τη νομική βάση ούτως ώστε να συμπεριληφθεί και το Κοινοβούλιο στη διαδικασία και έχουμε δύο νομικές βάσεις, την 167 και την 352 και επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η ιστορική συνείδηση. Έχουμε πάρει feedback, μια ανάδραση ας πούμε για αυτό το πράγμα που δείχνει ότι αυτό το σκέλος του προγράμματος είναι πολύ σημαντικό, αποδείχθηκε πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει αυτή η συνιστόσα της ιστορικής συνείδησης να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Τώρα, οι εμπλεκόμενοι στη βάση θα πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερο και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα, ε, πρέπει να δούμε επίσης και τι επίδραση έχουν και βραχυπρόθεσμα, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα ε, δούμε και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Όχι από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω προς τα πάνω θέλουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά και γι' αυτό η βάση είναι πολύ σημαντική. Ε, προκειμένου περί αυτών των προγραμμάτων και της πρόθεσής τους. Τώρα, για τον προϋπολογισμό, αυτό που προβλέπεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, που θα ελαχιστοποιηθεί, γιατί μόνο 30 εκατομμύρια το χρόνο ε, προβλέπονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά πρέπει λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε στους τομείς όπου θα είναι απαραίτητα. Και η Κομισιόν θα πρέπει να πάρει κάποια κονδύλια και για την επικοινωνία. Θα μπορούσε ίσως, να, αν θέλει χρήματα, να τα βρει από, άλλους, από άλλες πηγές, όχι από αυτά τα προγράμματα. Επίσης πρέπει να ληφθεί μέρη για την υπογράμμιση του ρόλου των αθλητικών οργανώσεων στην πρόταση. Και αν προχωρήσει το πρόγραμμα και κατανεμηθούν τα λίγα αυτά κονδύλια, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η κατανομή θα γίνει με τρόπο ίσο, να υπάρχει μια γεωγραφική ισορροπία στην κατανομή των πόρων. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Μετά, να σας πω ότι το Συμβούλιο ακόμη ε, δεν έχει εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό. Εκρεμεί στο Συμβούλιο η συζήτηση αυτή. Μάλλον τέλος Νοεμβρίου θα τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά με τον Φαν Ρόμπαϊ, αλλά Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει καλό δημοσιονομικό πλαίσιο και για αυτό το πρόγραμμα. Χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις, διότι ε, προωθούνται πολύ σημαντικά πράγματα. Και αν παίρνουμε μόνο 30 εκατομμύρια το χρόνο για να κατανεμηθούν, ε, δεν είναι ε, πολλά, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών. Και αν δούμε τώρα τα προτινόμενα κονδύλια, αυτά δεν φτάνουν ούτε στα, στο ύψος των κονδυλίων του τρέχοντος προγράμματος, ακόμα και όταν γίνει διόρθωση με βάση τον πληθωρισμό. Το μόνο πρόγραμμα σε ενωσιακό επίπεδο το οποίο προωθεί την ιστορική συνείδηση, την ιστορική μνήμη, είναι αυτό. Και αυτή η ιστορική μνήμη, η ιστορική συνείδηση θα οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις. Πρέπει λοιπόν να διατίθενται κονδύλια για να μιλήσουμε για τα αίτια του ολοκληρωτισμού και άλλα. Και πριν από πέντε χρόνια επίσης είχαμε αποφασίσει να μιλήσουμε για τον ναζισμό σταλινισμό και τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Είδαμε ότι και αυτά έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση και είναι θέματα που δίνουν έναυσμα για πολλές συζητήσεις. Η ιδέα είναι να δούμε, να πάμε πίσω στις ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, διασφαλίσουμε ότι τα δυσάρεστα και τα τραγικά δεν θα ξαναγίνουν στην Ευρώπη, όπως το ολοκαύτωμα κλπ. Και ότι ο, ο άνθρωπος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα την χάνουν σεβασμού τώρα και στο μέλλον. Ε, να πω επίσης και, και ορισμένα πράγματα για το ιστορικό στην ιστορία του προγράμματος. Δεν θα την παραθέσω τώρα, αλλά θα σας δείξω αυτό εδώ το φυλάδιο, το οποίο έλαβα με email και έχει διανεμηθεί και εδώ. Υπάρχει σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητα φυλάδιο και θέλω εδώ να συγχαρώ την Κομισιόν για την ε, δουλειά αυτή. Αναφέρει όλα τα σημαντικά. Όχι. Ναι, προς το, προς Κοινοβούλιο. Ναι, ναι, στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο. Καλά που το προσέξατε αυτό για να μην ευχαριστήσω τους λάθος ανθρώπους. Ναι. Κοίτα, ε, ε, πίσω προς την Κομισιόν, αλλά το Κοινοβούλιο εννοούσα. Ευχαριστούμε Κοινοβούλιο, συγχαρητήρια για την καλή δουλειά στους συντάκτες. Και τώρα είμαι έτοιμος να ακούσω τις δικές σας σκέψεις. Μετά από αυτά, να ευχαριστήσω και εγώ τους κυρίους και τις κυρίες που ανέλαβαν για λογαριασμό μας να κάνουν αυτή την ε, αυτό το φυλάδιο. Η κυρία Κώστα ε, είπε ότι καμιά φορά καθυστερεί, καθυστερούν όλα αυτά ε, και έρχονται όταν πάει να τελειώσει η έκθεση. Καλό είναι να γίνονται νωρίτερα. Αλλά η δουλειά ήταν εξαιρετική. Και πραγματικά ε, και εγώ Τη χρησιμοποιώ πολύ και πρέπει να σας συγχαρούμε και να σας χειροκροτήσουμε μάλιστα για τη δουλειά αυτή, η οποία είναι χρησιμότατη. Και ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ανοίγουμε τη συζήτηση. Ζαμπίνε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Χάνου Τάκουλα για την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο γενικότερα να ασχολούμεθα με ένα θέμα όπως αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα, παρόλο που από οικονομικής άποψης είναι από τα μικρότερα. Είναι σημαντικό γιατί απευθύνεται άμεσα στους πολίτες της Ένωσης, έναν προς έναν, στη βάση. Είναι η πρωτοβουλία grassroots, όπως τη λέμε τόσο ωραία, ε, η οποία δίνει ζωή στην Ευρώπη. Ε, δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε το πρόγραμμα αυτό γιατί αυτά που αποτελούν πρωτοβουλίες οργανώσεων βάσης πολλές φορές έχουν ε, βαθύτερο νόημα και μεγαλύτερο νόημα για τους πολίτες της Ευρώπης. Χαίρομαι γιατί ο Χάνου Τάκουλα μίλησε και για τις αδελφοποιήσεις των πόλεων, ε, γιατί σε όλη την ιστορία εξέλιξη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αδελφοποιήσεις πόλεων ήταν εκείνη η δυνατότητα που συνένωσε τον κόσμο. Ε, από την ε, ιστορία της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γίνεται αναφορά και στην βάση. Γι' αυτό χαίρομαι που αναδεικνύεται αυτή η πτυχή. μία μικρή ανησυχία που έχω και που με μικρές τροποποίησεις στο κείμενο μπορούμε να την διασκεδάσουμε είναι το θέμα της ε, κατάστασης ανταγωνισμού μεταξύ των πιθανών υποψηφίων και ετούντων για το πρόγραμμα αυτό ε, των μικρών ε, οργανώσεων που δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν. Ε, με ισοτιμία αντιμετωπίστηκαν στο σχέδιο της Κομισιόν τα πολλά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Οι μεγάλες οργανώσεις που έχουν πολλούς συνεργάτες και μπορούν να κάνουν πολλές προτάσεις αιτήσει να υπερισχύσουν των μικρών οργανώσεων και κινήσεων επιτοπίων. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν το πρόγραμμα να διατηρηθεί ως πρόγραμμα το οποίο στηρίζει τις επιτόπιες πρωτοβουλίες των πολιτών. Ε, έτσι συμβάλλει στην ευρωπαϊκή παιδεία με την ιστορική συνείδηση και με προσανατολισμό προς το μέλλον για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμβιώσουμε στο μέλλον, πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί, να καταλάβουμε ένα τον άλλον και να συνεργαζόμαστε. Είναι κρίμα που η Κομισιόν Ε, κράτησε το σε λίγα για την, ε, ε, τις εργασίες δημοσιότητας και εύχομαι να βελτιωθεί η κατάσταση γιατί όταν είναι τόσο μικρό το πρόγραμμα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί και την δημοσιότητα θα πρέπει όλα τα χρήματα να δίνονται στα προγράμματα ε, στον προϋπολογισμό, τώρα αν δούμε τον προϋπολογισμό τη δημοσιεύσεων της Κομισιόν, μπορούμε να βρούμε κάποιες ε, λύσεις για να μην χρηματοδοτεί ε, τις δημοσιεύσεις ο προϋπολογισμός αυτού του μικρού προγράμματος. καλό είναι να γίνουν διαβουλεύσεις και στο Κοινοβούλιο. Γιατί δηλαδή γιατί να μην ε, γίνουν διαβουλεύσει με το Κοινοβούλιο. Ε, υπήρχε τίποτα κρυφό, υπήρχε κάποιος λόγος για να μην ε, υπάρχει συναπόφαση. Μετά σκέφτηκα ότι μπορεί, μπορεί να υπήρχε κάτι κρυφό. ίσως να αυτό το θέμα των, των δημοσιεύσεων που έπρεπε να καλυφθούν από το πρόγραμμα. Να προσέξουμε τα λίγα λεφτά να πιάσουν τόπο. Θα χαιρόμουν πολύ αν ε, μπορούσαμε τουλάχιστον να ε, αυξήσουμε κατά τον, προϋπολογισμό, κατά τον ε, πληθωρισμό συγγνώμη, το πρόγραμμα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση για τη χρηματοοικονομική κρίση, τη συζήτηση για την Ευρώπη, που δείχνει τελευταία ότι γίνεται πολύ σημαντικό να συμμετέχουν πάντα οι άνθρωποι επί τόπου. Δεν μπορεί να τους ενημερώνουμε μόνο από πάνω προς τα κάτω. Θα πρέπει να αναπτυχθεί από τις βάσεις, από τις ρίζες της η Ευρώπη. Και γι' αυτό θα πρέπει να προοικοδοτηθεί καλύτερα το πρόγραμμα αυτό από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ναι, να, να, να, να βρούμε και τον Άγιο Βασίλειο, όμως να μας δώσει τα λεφτά. Κύριο Φίσας, πρώτα ευχαριστώ. Ως ε, Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Τάκουλα για το έργο που έκανε για την ε, ανοιχτή του διάθεση να συζητήσει με τι πολιτικέ ομάδε. Είχαμε μια συνεδρία σε σκιωδών στο Στρασβούργο, μείζονο ε, σημασία για να ανταλλάξουμε απόψει. Και παρατηρώ με χαρά ότι πολλέ τι προτάσει μα τι έλαβε υπόψη ε, στη γνωμοδότησή του εισηγητή. Όπω γνωρίζουμε, το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κεφάλαια. Ιστορική μνήμη, ευρωπαϊκή θα γίνει και ε, συμμετοχή των, ε, δημοκρατική συμμετοχή, συμμετοχή των πολιτών. Η δομή που προτείνει το Συμβούλιο που τροπεί σε ελαφρά ε, την, τη δομή και τα κεφάλαια, παρόλο αυτά είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε. Έπειτα η νομική βάση είναι αυτή που είναι καθώς πέρασε μετά από συνένεση ε, με τη δικασία της συναπόφασης και άρα ενισχύεται η ιστορική μνήμη. Η ιστορική μνήμη όχι για την ιστορία, αλλά για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Γι' αυτό έχει σημασία η ιστορική μνήμη, είναι ε, ένα δίδαγμα για το μέλλον. Επίσης βλέπω ότι ο κύριος Στάκουλα συμπεριέλαβε και κάποιες προτάσεις που κάναμε τη συνεδρία και όπως ε, στον αθλητισμό, τροπολογία 6 και τροπολογία 18 για τις τοπικές κοινωνίες. Συμφωνώ απόλυτα και με την Σαμπίν ότι όλα αυτά δεν πρέπει απλά να προάγουν ε, απλά τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να συνοδεύονται από συγκεκριμένε δράσεις, ώστε πραγματικά να δώσουμε όθηση στην Ευρώπη των πολιτών. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι το εργαλείο της αδελφοποίησης των πόλεων και πώς μπορούν να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές, οι τοπικοί φορείς σε αρκετές πτυχές αυτών των προγραμμάτων υπάρχουν πολλές προτάσεις. Δεν θέλουμε να πλημμυρίσουμε με τροφολογίες στον Κροτάκουλο που είσαι κάνει εξαιρετική δουλειά σε μια διαδικασία συνένεση με πολιτικές ε, ομάδες και μέσα στα πλαίσια οικονομικής ε, στενότητας που υπάρχει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κρίμα. Κρίμα, καθώς ένα πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Η Ευρώπη και τους πολίτες», δηλαδή είναι το πρόγραμμα που η Ευρώπη διαθέτει προς τη διάθεση των πολιτών της ε, να έχει τόσο ισχνά κονδύλια. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή η Ευρώπη δεν ε, λαμβάνει και τόσο σοβαρά υπόψη τους πολίτες της. Αυτό συμπερνεί κανεί. Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες αυτό τώρα. Ε, να ευχαριστήσω βεβαίως τον εισηγητή, τον κύριο Τάπλε, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, για τον τρόπο τον οποίο έθεσε το ζήτημα και όλες οι σχολείες που αντιμετώπισε ε, σε νομικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο, όπως ήδη ακούστηκε, να επισημάνουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι στην πραγματική διάθεση των τόσων πολλών ενώσεων, οργανώσεων, μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τον Ευρωπαίο πολίτη να κατανοήσει καλύτερα την Ευρώπη και το νόημά της, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την ταυτότητα της Ευρώπης, όπως και την ικανότητα που έχει να καταστεί τους ε, Ευρωπαίους πολίτες κοινωνούς αυτής της όλης ιδέας που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το έχω πει και άλλε φορέ, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό να συνοδευτεί από μια διοικητική απλούστευση ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ενώσεων, των οργανώσεων, των προσώπων και την συμμετοχή τους, δηλαδή δυνατότητα συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα και να ε, χρηματοδοτηθούν. Ε, είναι κάτι που να επισημάνουμε. Χρειάζεται μια απλοποίηση, γιατί συχνά μιλούμε για πολύ πολύ μικρούς φορείς ενώσεις που ζητούν συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε να υπάρχει ελευθερία συμμετοχή, είναι πολύ σημαντικό χωρί πολλέ φραγίδε, χωρί πολλή χορτούρα και πολλή γραφειοκρατία. Πριν από κάποιο διάστημα, ω ΕΛΚ, ε, είχαμε οργανώσει και μία ακρόαση για τα αλλοκληρωτικά καθεστώτα. Και υπήρξε αθρώα συμμετοχή, ιδίω από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δίπλα στην ε, πολύ ορθή και η υπενθύμηση του ολοκαυτώματος, καλό είναι να υπενθυμίσουμε και την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και την πορεία και την ιστορία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης διότι όλη αυτή η σύντηση για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα θα πρέπει να ειδωθεί αναλογικά και ισότιμα, καθώς η ευρωπαϊκή ιστορία είναι γεμάτη μαρτυρίες από όλες τις πλευρές. Δεν είναι μόνο το ολοκαύτωμα, αλλά και το δράμα που έζησαν πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ, Μάρκο. <clears throat> Ευχαριστώ, Μάρκο, κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ, Ντόρι. Να αναφερθώ κι εγώ σε κάποια πράγματα που ε, έθεσαν και οι προλαλήσαντες Το βασικό πρόγραμμα είναι προσφορά στις πολίτες να διαμορφώσουν κάτι. Αυτό είναι το βασικό. Να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους, ε, τις ιδέες τους, να μπορέσουν να τις βάλουν σε πράξη και ο προϋπολογισμός αυτό το σκοπό έχει, πόντος είναι μικρός. Ο βασικός, ο πιο σημαντικός ακόμα ε, ρόλος είναι να οικοδομήσουν από κάτω την Ευρώπη οι πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό τώρα με την κρίση που και με το διακυβερνητικό χαρακτήρα πολλών δράσεών μας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι απόλυτα κέρια σημασία γιατί δίνει επιτόπου στον κόσμο την δυνατότητα να βρίσκει επαφή ο ένας με τον άλλον και να εφαρμόζει ιδέες. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε και εμείς γιατί ε, ε, θα ήταν παράλογο οι εκλεγμένοι βουλευτές να μην έχουν λόγο, ειδικά για τη φύση αυτού του προγράμματος. Ξαναλέω, όπως είπαν κι άλλοι, αν ο προπολογισμό είναι τόσο μικρός θα πρέπει να διατίθεται επιτόπου με μικρά προγράμματα που θα έχουν πρωτοβουλίες, μικροί οργανισμοί που θα έχουν πρωτοβουλίες να μπορούν να αξιοποιούν τα κονδύλια. Η ιδέα της ευρωπαϊκής παιδείας από την άποψη της ιστορικής μνήμης και συνείδησης, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τον ολοκληρωτισμό των εθνικών σοσιαλισμών, πρέπει να μιλήσουμε και για το φασισμό και το σταλινισμό, γιατί και αυτό είναι κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Με όλους αυτούς τους ολοκληρωτισμούς θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε όσο διαφορετικοί και αν είναι ο ένας από τον άλλον για να οικοδομήσουμε καλύτερο οικοδομικό, ε, δημοκρατικό μέλλον. Παραμένει αυτό ευρωπαϊκό καθήκον και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι όπως και το θέμα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, της θρησκευτική ελευθερίας, της ανεξιθρησκείας, ε, της ελευθερίας από θρησκείες, και εδώ και ως προς αυτή την ε, πτυχή της καθημερινότητας στην Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει το πρόγραμμα, όπως και η ειρηνική συμβίωση ε, στην καθημερινότητα. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, μια και θα μπούμε στο καυτό θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα κοιτάξω κι εγώ να πω κάτι ώστε να ε, υπάρξουν ορισμένε αυξήσει, αν και έτσι όπω είναι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ, η κυρία Μπενεραπάτου. Merci, euh, Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως και οι συναδελφοί μου, έτσι και εγώ πιστεύω ότι το πνεύμα της έκθεσης αυτής επιβάλλει να έχουμε ένα σύστημα συναπόφασης. Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να βρισκόμαστε σε καθεστώς συναπόφασης. Για μένα το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική φάση της ιστορίας μας. Συζητάμε μια νέα συνθήκη. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση ανάμεσα σε εκλεγμένους εκπροσώπους και Ευρωπαίους πολιτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο περισσότερο τη νέα αυτή συνθήκη, επικοινωνώντα περισσότερο με του πολίτες. Πρέπει τα ζητήματα τα οποία συζητάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λαμβάνονται υπόψη και από τους Ευρωπαίους πολίτες, να κινητοποιούνται στου πολίτες. Πάρα πολλοί πολίτες θεωρούν ότι είμαστε πάρα πολύ απόμακροι. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε όλες αυτές τις δράσεις που θα εμπλέξουν περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τον προπολογισμό, συμφωνώ και εδώ με του συναδέλφου μου. Ο προβλεπόμενος προπολογισμό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν στο σύνολό του να προβλέπεται ένα συγκεκριμένο προπολογισμό για, τους, για συγκεκριμένε δράσει, για του φορεί δράση και για, τις, για την ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για συγκεκριμένε δράσει και δομέ. Πάλι τα πράγματα εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρα. Ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίση για μένα, τροπολογία παριθμών 8, όσον αφορά την μνήμη, την ιστορική μνήμη. Πολύπλοκο το ζήτημα αυτό και μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ στις συζητήσει που είχαμε. Όσον αφορά την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται εδώ πέρα ότι αναφερόμαστε μόνο στον σταλινισμό, στο ολοκαύτωμα θεωρώ ότι ξεχνάμε και αφήνουμε εκτός και άλλα προβλήματα όπως η απεικιοκρατία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή ιστορία εξαλείφοντας ή κρύβοντας την πολύ αυτή σημαντική διάσταση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Και αναφέρομαι στο φαινόμενο της απεικιοκρατίας. Εγώ είμαι Γαλλίδα και Αλγερινή. Θεωρώ ότι με γέννημα θρέμα της απεικιοκρατίας και αυτό το οποίο συζητάμε πάρα πολύ σήμερα και ιδίω στη Γαλλία είναι το θέμα του Ισλαμισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να συνδέσουμε τη συζήτηση αυτή με την απεικιοκρατία. Ότι η απεικιοκρατία διαμόρφωσε ολόκληρους πληθυσμούς οι οποίοι έχουν ασπαστεί το Ισλάμ και οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ε, έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας εντελώς διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά κυρίως τον, ε, τους, τον Ισλαμικό πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, ιδίως όσον αφορά την ιστορία της Αλγερίας, ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η επικρατή διαμόρφωσε πάρα πολύ την ιστορία της χώρας αυτής και κατ' επέκταση την ιστορία της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω το Χάνου Τάκουλα για την πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ λυπηρό ότι έγινε πια θέμα τεράστιο η νομική βάση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Τέσσερις σύντομες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρός και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γεωγραφική ισορροπία στην κατανομή των πόρων σε μεγαλύτερη ισορροπία από ό,τι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό δημιούργησε προβλήματα στο παρελθόν. Υπήρχαν προβλήματα εδώ δηλαδή. Τα κράτη-μέλη πρέπει όλα να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στο πρόγραμμα Γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά κόστη που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι δαπάνες. Εγώ είμαι από το βορρά και νομίζω ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα μπορεί να μας βοηθεί να βρίσκουμε μια ισορροπία. Μια η γεωγραφική ισορροπία, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό που θα μας τον ετοιμάσει η Κομισιόν. Εκείνη πρέπει να τον βρει. Επίσης, όλοι οι πολίτες, όλοι, μη, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν με τρόπο ισότιμο. Δεν θα στηρίζουμε δομές, θα στηρίζουμε προγράμματα προγράμματα που θα έχουν προκύψει από τη βάση. Ο κύριος Στάκουλα ακολουθεί το σωστό δρόμο σε αυτό το θέμα και είναι σημαντικό τα προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών να είναι προγράμματα που θα παρέχουν πληροφορίες στην μητρική γλώσσα κάθε φορά, στην κάθε χώρα. Ίσως ε, θα έπρεπε να υπάρχουν ε, σύνδεσμοι, πρόσωπα επαφής ε, σαν διαμεσολαβητές και αυτό επίσης απαιτεί πόρους και καλύτερη κατανομή των πόρων και εδώ. να ευχαριστήσω τέλος τον εισηγητή και να πω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό. Και Επίση να δούμε και το θέμα της νομικής βάσης, να το αποφασίσουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την ε, έκθεση Τάκουλα. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικές ε, οι δύο συνιστώσεις, ε, τώρα δηλαδή περιγράφονται πιο καλά από ό,τι στην αρχική πρόταση. Δεύτερον, ενισχύεται αυτή η δουλειά της μνήμης, της ιστορικής ε, μνήμης, εγώ ήμουν σε μια συνεδρίαση της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Ρωσία και δύο ώρες λέγαμε ότι τα σημερινά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας προκύπτουν από τη διαφορετική κατανόηση της ιστορίας. Εκεί οφείλονται. Οπότε έχει νόημα η πρόταση αυτή. Τρίτον, ε, ε, το είπε η κυρία Τρούπελ ήδη. Νομίζω, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, έχει νόημα με δεδομένο τον μικρό προϋπολογισμό να προωθηθούν μικρά προγράμματα. Και τέταρτη παρατήρηση που ανέφερε και ο κύριος ε, ε, Ράπος από την Φιλανδία, να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει που δεν να το αγνοήσουμε. Αυτά είναι, αυτές είναι οι θετικές παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Ε, τώρα, προβληματίζομαι λίγο με τα ποσοστά. Όχι ότι έχω αντίρρηση, αλλά προβληματίζομαι λίγο για το ιστορικό κομμάτι, για το κομμάτι της ιστορίας των πολιτών 20 προς 60%. Ίσως θα έπρεπε εδώ να υπάρχει κάποια δυνατότητα να το ξαναδούμε ή να το διαπραγματευτούμε. Μπορεί να τροποποιήσουμε λίγο τα ποσοστά, ούτω ώστε να αυξηθεί λιγάκι το ιστορικό κομμάτι. Αλλά θα τα ξαναπούμε αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση να κάνω κι εγώ. Οι υφιστάμενες δομές στον τομέα, ας πούμε το σπίτι της Ευρώπης, που είναι μεγάλος οργανισμός που συνενώνει ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν μεγάλη σημασία και είναι αναντικατάστατοι. Αν δεν ε, έχουν μια πάγια χρηματοδότηση θα μας λείψουν οι διαμεσολαβητές. Δεν ξέρω, Χάνου, υπάρχει δυσκολία στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτές οι ενδιάμεσες οργανώσεις που δρούν μεσολαβητικά δεν μπορούν να, να... χρηματοδοτούνται. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουν κάποια χρηματοδοτική υποστήριξη για τη δουλειά τους χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ε, ολόκληρη ιστορία και πολλές αιτήσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πάντα πίστευα ότι πριν από 12 χρόνια πριν από 14 χρόνια πίστευα ότι είχαμε πείσει την Κομισιόν ότι οι αιτήσει, τα έγγραφα αιτήσεων για την χρηματοδότηση αδελφοποιήσεων πόλεων θα έπρεπε να απλοποιηθούν και να είναι λιγότερο δαπανηρές. Γιατί δεν είναι και τεράστια τα ποσά που δίνονται για τις αδελφοποίησει. Εν τω μεταξύ όμως φαίνεται ότι ισχύει το αντίθετο. Γιατί μόνο στα λόγια άλλαξε κάτι, μου είπαν ότι ναι, ναι, ναι, κάναμε κάτι, αλλά οι άνθρωποι επιτόπου αντιμετωπίζουν μία θύελα, χαρτοθύελα ε, ε, ε γραφειοκρατική. Ε, δέστε το λοιπόν αυτό ε, για να ενημερωθεί και η Κομισιόν. Μου είπαν ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν, μια κυρία, μάλιστα κυρία μου, η κυρία Μπερνέτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ενώ γενικά στηρίζεται την ιδέα για αυτό το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020 και το σχέδιο του εισηγητή σας είναι γενικά θετικό έντε τις προτάσεις μας, τις προτάσεις μας και πράγματι ήδη το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε κάποιες α, τροποποιήσεις που προτείνει με τη γενική προσέγγιση που ακολουθεί προτάσεις που δεχθήκαμε καθώς βελτιώνουν την αρχική πρόταση γιατί την αλλάζουν και δεν αλλοιώνουν την αρχική φιλοσοφία της πρότασης. Πολλά στοιχεία στην ε, έκθεση του εισηγητή είναι θέματα που έχουμε ζητήσει και στο Συμβούλιο. Και θέλω να επισημάνω και κάποια από τα θέματα που ακούστηκαν σήμερα και συμπεριλαμβάνονται στην αναθεωρημένη πρόταση πλέον. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογή σχετικά με τη διάσταση της ε, ιστορικής μνήμης και της ηθαγένειας. Ο λόγος που συμπεριλαμβάνουμε αυτή τη διάσταση είναι για να κατανοήσουμε τις αιτίε των ακροτικών καθεστώτων στην Ευρώπη και να συμπεριλάβουμε και δράσεις που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης. Άρα δηλαδή ξεπερνούμε τα θέματα ναζισμού και σταλινισμού που κάναμε στο παρελθόν. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε δράσεις που είναι κατά της μυσαλλοδοξίας, της καλύτερης αλληλοκατανόησης, συνεννόησης και προσέγγισης για να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, όπως είπατε και εσείς οι ίδιοι. Κάτι που ήδη συζητήθηκε και λήφθη υπόψη από το Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα μικρά και τα μεγάλα project. Και αυτό γίνεται με τον εξή τρόπο. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να επιλέγουμε project που θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Κάτι άλλο που στήθηκε επί μακρόν στο Συμβούλιο και το λάβαμε υπόψη είναι η αρχή της γεωγραφικής διαφορετικότητας και δείτε στην ανθρωπίνη πρόταση εισαγάγαμε τέσσερις νέους δείκτες για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τη γεωγραφική διαφορετικότητα ε, του κάθε project. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και το διοικητικό κόστος, με χαρά θα σας παραπέμψω στην ε, έκθεση που σας έχουμε υποβάλει σε σύγκριση με προηγούμενα προγράμματα αυτή η πρόταση οδηγεί σε μια πολύ αποτελεσματική ε, της ε, δικαιωτικής διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές αιτήσει, το e-application, που είναι πολύ πιο εύκολος τρόπος υποβολής αίτησης για το παρελθόν. Επίσης χρησιμοποιούμε α, κατά πάγια, ε, ποσοστά ενιαίους συντελεστές και προσπαθούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε τεράστιες και χρονοβόρες διαδικασίες κατά την υποβολή της έντασης. Τώρα, για την επικοινωνία. Αν, αν θέλουμε να συμβάλλουμε στον τομέα της επικοινωνίας και της εταιρική επικοινωνίας συγκεκριμένα, τότε θα πρέπει να καταβάλουμε πιο στοχευμένες προσπάθειες χωρίς αναγκαστικά να πιέσουμε σε αύξηση του συνολικού προπολογισμού. Προτείναμε συγκεκριμένα σε όλες τις τομικές βάσεις να υπάρχει μια εξή ρήτρα. ότι ένα μέρος οποιοδήποτε πρόσθετο μπορεί, μπορεί λέω, και να ε, χρησιμοποιείται για την εταιρική επικοινωνία. Αυτό θα, με, θα αποφασίσετε συγγνώμη, με επιτροπολογία. Και άρα θα πηγαίνει στα κράτη-μέλη για να αποφασίσουν. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποια οικονομία κλίμακας και να εξοικονομήσουμε πόρους. Αυτό είναι η εταιρική επικοινωνία. Αυτό να μην το μπερδέψουμε με την αξιοποίηση, που είναι μια άλλη έννοια προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσω της πρότασης, μέσω της επανεξέτασης ομοτήμων, τα peer reviews, να μπορούμε από κοινού όλοι μαζί να επιλέγουμε τα καλύτερα project με βάση τις καλές πρακτικές. Και αυτό που βεβαίω μένει και είναι στοιχείο κλειδί είναι νομική βάση, το άφησα για το τέλος, προς το παρόν η θέση μας παραμένει ίδια. Η ανάλυση που έκανε η νομική υπηρεσία διαφέρει από την ανάλυση που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι η πρόταση μπορεί να βασιστεί μόνο στο άρθρο 352 και διπλή νομική βάση ούτως ή άλλως για νομικούς λόγους δεν είναι εφικτή διότι οι δικασίες υιοθέτησης δεν είναι συμβατές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τώρα πλέον συζητάτε την πρόταση στην ουσία της και αυτό μας ενθαρρύνει, θεωρούμε ότι επί της ουσίας οι θέσεις μας δεν διαφέρουν σημαντικά και μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα απάντηση για οργανισμούς όπως το σπίτι της Ευρώπης. Κομισιόν πάλι. Ναι, σας ζητώ συγγνώμη. Όντως, το νέο προβλεπόμενο πρόγραμμα προβλέπονται επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις πολυετής. Επομένως, θα υλοποιηθεί η χρηματοδότηση αυτή, εφόσον υπάρχει όμως και αντίστοιχη πρόταση. Η δομή πάντω η οποία υφίσταται για το νυν πρόγραμμα πρόκειται να επανληφθεί και για το μελλοντικό πρόγραμμα, επομένω θα προβλέπεται χρηματοδότηση και για τι δομέ αυτέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα τώρα πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες προτάσεις και παραμβάσεις σας. Τόσα ευχαριστώ ακούστηκαν που πρέπει να προσθέσω και εγώ τα, τα δικά μου ε, σε όσους συνεργάστηκαν μαζί μου, γιατί πρόκειται για συνεργατική δουλειά. Τώρα, για τον προϋπολογισμό, είναι επί του παρόντος δύσκολο να πούμε κάτι, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό οριστικό ποσό. Γι' αυτό μιλάμε μόνο για ποσοστά, όπως και στις εκθέσεις της Προέδρου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι δικές μου οι προτάσεις πάνε προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου, δηλαδή 60% για τις αδελφοποίησεις και τις σχετικές δραστηριότητες, 25% ιστορική συνείδηση, λίγο παραπάνω δηλαδή από την πρόταση που έχει γίνει, του 20%, διοίκηση 10% και οριζόντιες δραστηριότητες 20% επίσης. Τώρα, για τον προϋπολογισμό, συμφωνώ απόλυτα με τον Μάρκο όταν λέει ότι αυτό είναι πραγματικά πρόγραμμα των πολιτών, των Ευρωπαίων και είναι πολύ οδυνηρό ότι ο προϋπολογισμός είναι τόσο μικρός, λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια. Κάτι λέει όμως και αυτό. Στην προηγούμενη εκλογική περίοδο 400 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό πήγαν στη καλλιέργεια καπνού. Παράδειγμα. Ενώ λέμε τόσα και τόσα για την επικινδυνότητα του καπνίσματος. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν είναι πάντοτε ισορροπημένη η πολιτική μας και αυτό συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Είναι και ένα πρόβλημα αν θέλετε νομιμοποίησης γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι η Ένωση δεν είναι για αυτούς εκεί δεν τους εξυπηρετεί. Γι' αυτό είναι το πρόγραμμα σημαντικό, γιατί είναι πρόγραμμα των πολιτών, είναι πρόγραμμα της βάσης. Ευχαριστώ θερμά και την Κομισιόν, σε μεγάλο βαθμό ομονοούμε, αλλά η νομική βάση ε, είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι καλό είναι να προσεγγίσετε λίγο τη δική μας τη θέση. Τέλος πάντων, θα οψόμεθα. Τι αποτελέσματα θα ε, έχουμε και από εκεί. Πάντως, ε, ε προς το παρόν είναι σημαντικό να πούμε ότι μέχρι τις 24... Α, ε, ε, η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών είναι 24 Οκτωβρίου και σήμερα στη συνεδρίαση των συντονιστών θα τα ξαναπούμε αυτά. Πάντως θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα με βάση τη διαδικασία συναπόφασης και ελπίζουμε ότι στην Ευρώπη των πολιτών θα μπορούν να ε, συμμετέχουν οι πολίτες όντως και η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα συμβάλλουν στη δημιουργία καλής βάσης και καλού προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ε, συνεισφορές σας. Και ελπίζω ότι τα κατέγραψα όλα όσα είπατε. Να προσθέσω κάτι μην κατηγορούμε μόνο. Έχουμε το πρόγραμμα για την ιδιότητα του πολίτη, το citizenship, αλλά και τα άλλα προγράμματα για τον πολίτη είναι και αυτά. Για, το, για τους πολίτες, το πολιτιστικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό δεν είναι για μας, ούτε για κάποιους ε, ε, ψηλό βαθμούς που δεν ενδιαφέρονται. Όλα αυτά είναι για τους πολίτες που με ενσυναίσθηση θα συμβάλλουν στην Ευρώπη που τους ανήκει. Γιατί αν ε, ε, η Ευρώπη δεν εξελιχθεί σωστά θα ζημιώσουν όλοι. Αλήθεια είναι, δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για το πρόγραμμα αυτό, αλλά ε, πόσο μάλλον θα, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, αυτά που υπάρχουν. Έχεις δίκιο εκεί. Είπες για την καλλιέργεια του καπνού. Ο καπνός που στηρίζεται δεν καπνίζεται. Αυτός είναι βιομηχανικός καπνός για βιομηχανική χρήση. Καπνός υπάρχει και στα τραπεζογραμμάτια. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε υπερβολικοί. Και εγώ το κάνω. Ε, υπάρχουν καπνεργάτες που δουλεύουν, που αλλιώς θα χάσουν τη δουλειά τους. Μην κάνουμε λοιπόν τέτοιες συγκρίσεις. Δεν είναι καπνός αυτός που, που ε, επιδοτείται, δεν είναι καπνός για να τον καπνίζουμε. Ωραία, είπε 24 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών και 26-27 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της επίσημης ημερησίας διάταξης. Όσοι δεν είναι συντονιστές ας εγκαταλείψουν την ωραία αυτή αίθουσα. Καλό σας βράδυ. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε ακόμα, όμως χωρίς τη δική σας παρουσία.